Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών. Εγώ θα προεδρεύσω αυτό το απόγευμα. Λίγες ανακοινώσεις πριν περάσουμε στην ακρόαση. Καταρχήν μπορούμε να εγκρίνουμε την ημέρηση διάταξη. Συμφωνείτε έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων της 21ης Μαρτίου και 27ης Μαρτίου 2017. Εγκρίνονται πολύ ωραία. Ανακοινώσεις Προέδρου δεν υπάρχουν από ό,τι ξέρω και γι' αυτό περάσουμε στην ακρόαση. Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που είναι μαζί μας η Μέρι Ρόμπινσον πρόεδρος της Ιρλανδίας από το 1990 μέχρι το 1997 και πρόεδρος του Ιδρύματος Μέρι Ρόμπινσον για την κλιματική δικαιοσύνη. Θα μας κάνει την εισαγωγική ομιλία για την κλιματική δικαιοσύνη και χωρίς άλλη χρονότριβη να δώσω το λόγο στην Μέρι Ρόμπινσον. ένα διαδικαστικό από τον κύριο Ταραπέλα. Τρέχω ιδιαίτερο σεβασμό και θαυμασμό προς την κυρία Ρόμπινσον. Μάλιστα τη γνώρισα ε, όταν διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα θεσμικά όργανα, πριν το πολύ σημαντικό ρόλο που ανέβαλε και στην ε, Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Χθες ε, όλοι μάθαμε ότι η Σαντική Αραβία ορίστηκε μέλο τη Επιτροπή Γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη. Εμείναμε ευρώντη παγκοσμίω με την ειδησία αυτή. Δηλαδή, υποτίθεται ότι η Σαουδική Αραβία θα προωθήσει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών στον κόσμο. Ε, θα μπορούσε να προκαλέσει μηδίαμα, ε, αν δεν ήταν τόσο τραγελαφικό και σκανδαλώδε. Η Σαουδική Αραβία θεωρεί υποδέστερε τι γυναίκε καθ' τη διάρκεια τη ζωή του και τη μόνιμη κυδαιμονία των ανδρών. Απαγορεύεται μάλιστα στι γυναίκε να οδηγούν αυτοκίνητο στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα το Μάρτιο ε, εγγενίασε ένα συμβούλιο για τις γυναίκες ε, χωρίς ούτε ένα μέρος γυναίκες. Ε, γενιοφόροι άνδρες μόνο προεδρεύουν στο συμβούλιο αυτό. Βέβαια έγινε τεράστιο λόμπι από τη Σαουδική Αραβία για να λάβει αυτή τη θέση ε, στα Ηνωμένα Έθνη με μοναδικό ενδιαφέρον ή συμφέρον να πάρει αυτό το σήμα το, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκέ χώρε ψήφισαν υπέρ τη συμμετοχή τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Έθνη. Έγιναν συνένοχοι αυτού του τραγέλαφου. Είναι νιωστή η παραβίαση που κάνει στα δικαιώματα των γυναικών η Σαουδική Αραβία και νιώθω καθήκον ω μέλο τη Επιτροπή Γυναικών να καταγγείλω και να στυλιτεύσω αυτή την κατάσταση μια και δεν είναι της παρούσης της σημερινής ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την γελιότητα, αυτή, αυτό το τραγέλαφο που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη, αυτή την κοροϊδία, γιατί πραγματικά είναι προσβολή ύβρις προς τις γυναίκες ε, και θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτή την κατάσταση. Και πρόκειται για ένα ψευτοσύμμαχο, για μια χώρα που προωθεί ε, παρόλα αυτά έναν ε, ε, φανατικό Ισλαμισμό, εξτρεμιστικό και ακραίο και νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και ίσως και ε, στην Ολομέλεια δεν μπορούμε να, περάσουμε, να αφήσουμε να περάσει στον Ντούκου αυτή η κοροϊδία, αυτός ο τραγέλαφος με τη συμμετοχή της ε, Σαουδικής Αραβίας στα Ηνωμένα Έθνη στην Επιτροπή για τις Γυναίκες. Λυπούμε που διατάραξα κάπως την ομαλή διεξαγωγή της δημόσιας ακρόσης. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Ναι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί σας και θα το θέσουμε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, πώς θα ενεργήσουμε. Φαντάζομαι ότι ε, όλοι συμφωνούμε και στενιζόμαστε τα σχόλιά σας για το θέμα αυτό. Πριν δώσω το λόγο στη Μέρη Ρόμπινσον, καλύτερα σας δώσω το λόγο στην κυρία Άμστραμ, που είναι η συγκήτριά μας για την κλιματική δικαιοσύνη. Γνωρίζω ότι περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία την ομιλία της Μέρι Ρόμπινς και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που είναι παρούσα εδώ στην ακρόαση μας σήμερα. Εγώ θα κάνω κάποια σύντομα εισαγωγικά σχόλια, ξεκινώντας ε, καταρχήν με ένα θερμό καλωσόρισμα προς τους καλεσμένους, τους εμπειρογνώμονες, ε, όλους ε, τους παρόντες. Για μένα τουλάχιστον η Μέρι Ρόμπινσον ενσαρκώνει τον αγώνα για την κλιματική δικαιοσύνη από πολιτική άποψη και ε, υψώνει τη φωνή των εκατομμυρίων ανδρών και γυναικών που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε παγκόσμια δικαιοσύνη για αυτούς, ε, τους ξεχασμένους ανθρώπους, ε, γιατί είναι περιθωριοποιημένοι, αποκλεισμένοι και ξεχασμένοι. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς όλοι και οι επερχόμενες γενιές να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν δράσουμε τώρα θα βρεθούμε όλοι χαμένοι. Επίση χαίρομαι για την παρουσία τη Τζάνι Στεφανσό και τη Στεφάνια Λαζότο, γιατί πρόκειται για ακτιβίστριε που είναι μάρτυρες της κλιματικής αλλαγής που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή και που μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους. Θα πρέπει να μας συμβουλεύσουν πώς μπορούμε και εμείς ως πολιτικοί να προχωρήσουμε. Και η ιστορική συμφωνία των Παρισίων τη περασμένη χρονιά είναι πραγματικά μια ρηξικέλευτη πρόοδο που θα προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών κατά την ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων. Επίση, τάσεται υπέρ τη δημιουργία ικανοτήτων για τι γυναίκε και την λήψη υπόψη τη διάσταση του φύλου. Γιατί οι κλιματικέ αλλαγέ επηρεάζουν δυσμενώ και τα κορίτσια και τι γυναίκε και μάλιστα οξύνουν τις υπάρχουσες ε, ανισότητες, τις διακρίσεις, ε, την ενδοκοικογενειακή βία που βιώνουν καθημερινά πολλές γυναίκες. Και νομίζω ότι ε, Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκε πρωτοστάτησαν στι προσπάθειε μετριασμού, ήταν καταπληκτικέ ακτιβίστριε στι κοινότητέ του, στι οικογένειέ του, στι οικονομίε του και συνέβαλαν στην καταπολέμηση των ακραίων ε, αποτελεσμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα. Και μάλιστα ήταν υπέρ ε, πρωτοβουλειών χωρί αποκλεισμού. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του στην διαδικασία λήξη αποφάσεων δεν είναι επαρκή, ούτε λαμβάνονται ε, δεόντως ε, τα συμφέροντα τους ε, και τα δικαιώματά τους στα διάφορα σχέδια δράσης και απειλούνται με περισσότερες ανισότητες και αποκλεισμό. Και μάλιστα η ελληπή συμμετοχή του στην τελική σύλληψη αποφάσεων ευθυνόταν και για το χαμηλό βαθμό προόδου των κλιματικών στρατηγικών και πολιτικών μας. Μάλιστα και παρόλο που το σχετικό ταμείο τάχθηκε υπέρ της των φύλων. Τα κονδύλια για τις περιβαλλοντικές δράσεις ελάχιστα εξασφαλίζουν ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση για προγράμματα που έχουν τις γυναίκες ως διαχειρίστριες ή ως δικαιούχος. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν και το Ταμείο για το Περιβάλλον και το Ταμείο για την Πράσινη Ανάπτυξη να ενισχύσει τα κονδύλια για ειδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση μιας δικαιοσύνης κλιματικής αλλά και της ισότητας των φύλων. Και την επιτακτική ανάγκη αυτή η δράση. Το 2015 η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε έκθεση που δείχνει ότι οι κλιματικές αλλαγές σε περιοχές όπως η Ποσαχάριος Αφρική και η Νότια Ασία μπορεί να εξαναγκάσει έως και 100 εκατομμύρια ανθρώπους ε, σε εξαθλίωση μέχρι το 2030 και χωρίς ακριβωδή και η κατανομή των πόρων θα έχουμε εκατομμύρια εκτοπιστέντε ε, για περιβαλλοντικούς λόγους. Μάλιστα τα Ηνωμένα Εθνή υπολογίζουν ότι ε, μέχρι το 2050 έχουμε και 200 εκατομμύρια περιβαλλοντικού πρόσφυγε. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε το σχετικό θεματολόγιο για να προσαρμόσουμε ε, τις κλιματικές, να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να αποφύγουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες. Έχουμε μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να ε, χρησιμοποιήσουμε τις κλιματικές δράσεις για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και να κάνουμε ακουστή τη φωνή των κορισιών και των γυναικών. Να τι φέρουμε στο επίκεντρο όλων των κλιματικών περιβαλλοντικών προσπαθειών και των σχετικών επενδύσεων. Επίση, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία τη έκθεση που θα απευθύνουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για το πώ μπορούμε να αναπτύξουμε στρατηγικέ, να προωθήσουμε περαιτέρω την ισότητα των φύλων σε ένα πλαίσιο κλιματική δικαιοσύνη γιατί ζούμε σε ένα σταθές πολιτικό περιβάλλον. Ε, έχουμε τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Brexit, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά τα θέματα της κλιματικής δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων ε, είναι θέματα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα ε, παραμερίζουμε ή να τα κρύβουμε πίσω από ένα παραπέτασμα καπνού. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στη συζήτηση και να ανταλλάξουμε υπόψη Και χαίρομαι για την διεξαγωγή αυτής της δημοσιακρόασης. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητρία. Και τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, δίνω το λόγο στην τέωσα πρώτη τη την κυρία Μέρι Ρόμπινσον, που είναι πρόεδρος τώρα του Ιδρύματος Μέρι Ρόμπινσον. Μεγάλη τιμή μας να είστε μαζί μας σήμερα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια Λίνα Εγκστρώμα και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση, διότι είναι πράγματι σημαντική έκθεση αλλά και η ακρόαση σε ό,τι αφορά την ισότητα των φίλων και την κλιματική δικαιοσύνη για τον ρόλο των γυναικών. Χαίρομαι που έχω προσκληθεί εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορώ να συμμετέχω στη σημερινή αυτή ακρόαση. Θα εστιάσω σε θέματα πολύ προσφυλή για μένα που είναι οι γυναίκε, ε, κλιματική δικαιοσύνη και η ισότητα των φίλων. Χρειαζόμαστε την Επιτροπή των Γυναικών αλλά και τι άλλε επιτροπέ του Κοινοβουλίου ώστε να φροντίσουν ότι οι γυναίκε, κλιματική δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων είναι κομβικά θέματα ε, σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή τη ε, συνθήκη των Παρισιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά συνεχίζουμε να υποτιμούμε τη διάσταση του φύλου ε, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, παρά τα όσα γίνονται σε επίπεδο ΟΗΕ, για να υπάρχει μια ατζέντα, ένα θεματολόγιο για την ισότητα και τα δικά μάτια μπορώ να πω ότι άνοιξαν πέρυσι, οπότε και ταξίδεψα στι χώρε που πλήττονται ιδιαίτερα από τη κλιματική αλλαγή ως ειδική απεσταλμένη ε, του ΟΗΕ για το Ελνίνιο και το κλίμα και εκεί πραγματικά είδα την τρομερή ξηρασία που προκαλεί το φαινόμενο Ελνίνιο. Επισκέφθηκα την Ονδούρα επίσης ε, ε, στον στεγνό διάδρομο της Κεντρικής Αμερικής πήγα που είδα πόσο πλήττεται επίσης από το φαινόμενο Ελνίνιο και πραγματικά αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα διότι οι τοπικές κοινωνίες είχαν ήδη εξασθενήσει με, τις, ε, με τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Συνάντησα γυναίκες από διάφορα τοπικά ε, χωριά στο πλαίσιο μιας ΜΚΟ. Κάθισα κάτω από ένα ε, δέντρο και είδα και άκουσα, είδα τον πόνο στα πρόσωπά τους. Μια γυναίκα με ρώτησε πώς ζείτε χωρίς νερό. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω. Πώς μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς νερό. Αυτό ήταν το ερώτημα μου είπαν τα προβλήματά του αυτέ οι γυναίκε, αλλά μετά μου είπαν ότι είναι αποφασισμένε, θέλουν να έχουν μεγαλύτερη αθεκτικότητα αντοχή, να φροντίσουν για την μερία του χωριού. Και πήγαιναν με κουβάδε και μάζευαν νερό, ε, δηλαδή τροφοδοτούσαν τα χωριά του με νερό. Επίση, ε, καλλιεργούσαν διάφορα φυτά, γιατί είδαν ότι το, ο αραβόστο δεν είναι ένα καλό φυτό, δεν ευδοκιμεί σε συνθήκε ξηρασία και καλλιεργούσαν πιο αθεκτικά λαχανικά φυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα εδώ. Γυναίκε επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την κλιματική αλλαγή λόγω των παραδοσιακών ρόλων που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Δεν είναι όμω μόνο θύματα, όλο και περισσότερο είναι οι φορεί αλλαγών. Εμεί στο Ίδρυμά μου στηρίζουμε τη σημασία που έχει το να συμμετέχουν οι απλέ γυναίκε. Οι παραδοσιακέ γνώσει του είναι πάρα πολύ χρήσιμε στην όλη προσπάθεια ήθελα να ακούσω και τι έχει να πει το Συμβούλιο ΣΑΜΗ και οι συνάδελφοι που είναι εδώ από αυτό το οργανισμό για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να θυμόμαστε πόσο δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, εφαρμογή της συνθήκης των Παρισίων. Ότι θα σέβεται, θα προάγει ε, και θα εφαρμόζει τις ε, υποχρεώσεις και για την ισότητα των φύλων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κλιματική δικαιοσύνη. Η κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερη ανισότητα. Είναι άνηση η κλιματική αλλαγή και αυτό σημαίνει ότι οι πλέον ευάλωτοι είναι και αυτοί που μάλιστα έχουν ε, λιγότερο, λιγότερη ευθύνη, αλλά αυτοί θα ε, πληγούν περισσότερο με 1,5 βαθμό Κελσίου παραπάνω ε, αλλάζει ο κόσμος ε, για πάντα, για πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Θέλουμε την κλιματική δίκαιωση να τη βάλουμε στο επίκεντρο της κλιματικής δράσης. Ζητούμε λοιπόν μεγαλύτερη φιλοδοξία από τις χώρες ε, για να μειώσουν τις εκπομπές οξυδίου του άνθρακα και να προστατεύσουν τους πολίτες από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα θυμάστε ότι στην προετοιμασία της διάσκεψης αυτής των Παρισίων έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το η Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με άλλες ε, ε, Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πει ότι τουλάχιστον το 20% του προπολογισμού μέχρι το 2020, 180 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, θα διατεθούν για τι δράσει που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματο, όπω είναι τριασμό τη αλλαγή του κλίματος, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματο. Δείχνει αυτό πόσο ε, προσιλωμένη είναι στο να προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του πολίτε από τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή και να επενδύσει στι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια για το μέλλον. όπω γνωρίζουμε, κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο μόνο του ε, κατοικού των ψωμένων χωρών, αλλά και τι κοινωνίε εδώ, εμά, ε, στην Ευρώπη. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν όλο και πιο όλο και πιο σοβαρά. Διάφορε περιφέρειε στην Ευρώπη θα έχουν ε, ίσω διαφορετικά, θα πληγούν διαφορετικά και ίσω και ανάλογα, διαφορετικά θα πληγούν και τα διάφορα στρώματα τη κοινωνία και αν ισομερώσει. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Θέλουμε να αναπτύξουμε πολιτικέ και να κάνουμε ενέργειε οι οποίε θα είναι μετασχηματιστικές και θα φέρουν ισοτιμία. Συμμετοχή, διαφάνεια, λογοδοσία. Αυτές είναι οι βασικές αρχές ε, και θα εστιάσω πρώτα απ' όλα στη συμμετοχή. Αν θέλουμε να εφαρμοστεί ισότιμα, δίκαια και από όλου ε, ε, η Συμφωνία των Παρισίων, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να ακουστούν οι φωνέ αυτών που δυσανάλογα πλήττονται. Επίση, πρέπει να έχουμε ανταλλαγή γνώσεων ε, για την αντιμετώπιση των του κλίματο. πρέπει να μάθουμε από είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου και να δράσουμε αναλόγω. Και οι φωνέ των γυναικών πρέπει να ακουστούν ε, στο πλαίσιο τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι και το ε, πιο ευφυέ που μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι και το πιο σκόπιμο και αποτελεσματικό. Έχουμε πάρει απόψει από τι γυναίκε για την έκθεσή μα The Full View, για γυναίκες, από γυναίκε που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και είδαμε πόσο θετική είναι η συνεισφορά κράτους οι γυναίκες όπως ε, μια ε, γυναίκα μια παιδιά στο κεντρικό Βιετνάμ και άλλες αγρότησες που έχουν πληγεί εκεί λόγω καταιγίδων ε, έντονων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. Έχει κάνει πάρα πολλά. Η Ράνη συγκεκριμένη αυτή η Βιετναμέζα, συμμετείχε σε ένα project σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την κυβέρνηση του Βιετνάμ για τη μεγαλύτερη αντοχή των γυναικών και των τοπικών κοινωνιών σε ακρά καιρικά φαινόμενα. είπε και η Ιράν ότι χάρη στην καλή προετοιμασία κανείς στο χωριό δεν είχε στη ζωή του ούτε τραυματίστηκε στις καταιγίδες της περσινής χρονιά. Και η ιστορία αυτή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούμε στην αλλαγή του κλίματος. Ε, οι γυναίκες αυτές, οι αγρότησες, ε, τους δόθηκε ευκαιρία να βρουν ε, τρόπους να αντιμετωπίσουν, να είναι πιο ανθεκτικές στις αλλαγές του κλίματος. Στόχος είναι λοιπόν να εντοπίσουμε, να προβληματιστούμε και να ορίσουμε παρεμβάσει για να αντιμετωπίσουμε και κάποιε μεροληψίε που έχουν να κάνουν με το φύλλο και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει στη φάση τη υλοποίηση τη Συμφωνία των Παρισίων να δημιουργήσει ε, το πλαίσιο για μια υπεύθυνη κλιματική δράση και πολιτική. Να εστιάσω σε μία πτυχή. Έχουμε το σχέδιο δράσης ε, τρίπλη ε, C ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε στη δική της συνεισφορά ότι ανάγκη είναι να υπάρξει περισσότερη δράση για την ισότητα των φύλων, για τη χειραφέτηση αδρών, ε, για συγγνώμη, γυναικών και ε, κοριτσιών. Είναι μια πολύ καλή πρόθεση και καλό είναι να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και να δημιουργήσει ε, τις συνθήκες για την αντιμετώπιση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η έκθεση Full View του Ιδρύματός μας εντοπίζει συγκεκριμένα βήματα μπορούν να κάνουν όλοι οι μπλεκόμενοι φορείς για να επιταχύνουν την πρόοδο προ την ε, ισορροπία μεταξύ των φύλων. Υπάρχουν συστάσει όπως να έχουμε κάποιους ε, στόχους εκθετικής αύξησης, αποζημίωση οδηπορικών, δημιουργία ενός δικτύου, ισότητας των φύλων κτλ. Το δικαίωμα στη συμμετοχή μπορεί και Ένωση να το υποστηρίξει ώστε οι γυναίκε να μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσει ε, στο πλαίσιο του GNF να δημιουργηθεί ένα φόρουμ για όλους αυτούς ε, τους φορείς και για τις απλές γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν. Θα πρέπει οι διαπραγματεύτες και απλές γυναίκες να έχουν πραγματική επικοινωνία γιατί έχουν γυναίκε γνώσει που μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν και να έχουν μια πολύ ενεργό συμμετοχή. Πρέπει να στηρίξουμε τι γυναίκε αυτέ και τι δυνατότητε να μπορούν να μιλούν, να εκπροσωπούν τι ε, τοπικέ κοινωνίε και να τονίζουν τι προτεραιότητε. Εξίσου σημαντικό όμω είναι και τα μέλη του Ευρωπαϊκού και οι συμμετέχοντε ε, στο UNFCCC να ακούν τι γυναίκε πραγματικά. Όχι απλά να ακούνε κάτι, ότι κάτι λένε αυτέ οι γυναίκε, αλλά να προσέχουν πραγματικά τι λένε αυτέ οι γυναίκε. Επίση, σε λογοδοσία και διαφάνεια. Φαίνεται ότι αν υπάρχει διαβούλευση, συνεννόηση και αν συμμετέχουν ε, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορεί ε, στη δικασία λήψη αποφάσεων, ε, θα είναι πιο επιτυχημένε και αποτελεσματικέ οι δράσει. Δυστυχώ, μειώνεται η βάση αυτή τη στιγμή σε το κοινό των πολιτών. Υπάρχει καταστολή, συρρήγνωση. Υπάρχουν όμω οργανώσει που προσπαθούν να υποστηρίξουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά δικαιώματα, τη δημοκρατία. Θα πρέπει αυτό το σημαντικό χώρο να τον προστατεύσουμε στην κοινωνία μα και στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό φορέα ε, η ε, κοινωνία των πολιτών. Αυτή είναι η λύση κατά την άποψή μου και για την αντιμετώπιση της ε, αλλαγής του κλίματος και εσείς ελπίζω και εγώ ήμουν ε, σε μια ε, πορεία υπέρ της ειρήνης όπως έγινε στο Δουβλίνο αλλά και σε άλλες, της επιστήμης συγγνώμη. Και σίγουρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία και βλέπουμε ότι υπάρχουν οι τρόποι κινητοποίησης αυτοί που έχουν την θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και αν ακούσουν ε, κάποιες ε, φωνές αντιφρονούντων ε, θα αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που θα τους κάνουν πιο ισχυρούς ηγέτες. Θα πρέπει τα δικαιώματα των ανθρώπων να μπουν στο επίκεντρο της εφαρμογής συμφωνίας των Παρισίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει δύναμη στις φωνές που πολλές φορές δεν ακούγονται θα είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητά μα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαστε στο επίκεντρο ε, στον αγώνα κατά τη κλιματική αλλαγή. Ε, και οι γυναίκε δεν είναι θύματα, αλλά είναι φορεί αλλαγή. Οι γυναίκε πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη πηγαίνουν χέρι-χέρι για να έχουμε ένα μέλλον όπω αυτό που επιθυμούμε και θέλουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε ε, στένος και από τα λόγια του δεσμότητα του Ντέσμον οποίο μου είχε πει ε, όταν ήμασταν σε ένα πάνελ στη Νέα Υόρκη πριν από 6-7 χρόνια, κάτι που μου έμεινε, ε, κάτι που δεν θα ξεχάσω, ήταν μια κοινωνική σύναξη ε, πολλών ε, νεαρών που ήταν μπροστά στις ταμπλέτες τους και μέσω Twitter είχαν επικοινωνία και ήταν ενθουσιασμένος ο Ντεσμοντού, του το έδειχνε και με τις κινήσεις του, πόσο χαίρεται. Ο συντονιστής του είπε κάπως απότομα ε, γιατί είστε τόσο αισιόδοξο και ήταν γυναίκα η συντονίστρα και την κοίταξε και τη είπε, Όχι, Ντύρι, δεν είμαι αισιόδοξο. Είμαι φυλακισμένο τη ελπίδα, κρατούμενο τη ελπίδα. Prisoner of hope. Και είναι κάτι πολύ δυνατό ω έκφραση. Η ελπίδα σου δίνει δράση, σου δίνει ενέργεια, σου δίνει χώρο για να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να μην μπορεί ε, να τα λύσει όλα. Ε, μπορεί να είναι μισογεμάτο το ποτήρι, αλλά σίγουρα είναι αρκετά γεμάτο για να μπορεί να προχωρήσει, ε, να ενεργοποιηθεί και αυτό κάνει και η δική σα επιτροπή. Και η ισότητα των φίλων και η κλιματική δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε όλοι φυλακισμένοι τη ελπίδα, κρατούμενοι τη ελπίδα και να προωθήσουμε την ισότητα των φίλων και την κλιματική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μας δώσατε πολύ τροφή για σκέψη ε, και μας εμπνεύσατε με αυτά που μας είπατε. Ε, αλλά θα πρέπει η ακρόαση να συνεχίσει και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ελίνα Μπάντραμ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επικεφαλής της μονάδας Α1 που ασχολείται με διεθνείς ε, και διοργανικές σχέσεις στην Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Η κυρία Μπάρτεν θα πρέπει να φύγει γύρω στις 5, αλλά οπωσδήποτε οι συνάδελφός της, η κυρία Καρίνη Γκέντη, η οποία είναι ε, αναπληρωτής ε, διευθύντρια στην ε, μονάδα C1 Κλιματική Αλλαγή, θα μείνει μαζί μας. Η κυρία Μπαρνταράμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω την δυνατότητα να πάρω το λόγο ενώπιόν σας μετά από μια τόσο έγκριτη ομιλήτρια που γνωρίζουμε ότι έχει κάνει τόσα πράγματα, έχει πετύχει πετύχει τόσα πολλά ε, και στα πλαίσια της UNFC ε, ε, αλλά και γενικότερα όσον αφορά την δικαιοσύνη και την ισότητα των φίλων. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά εμπνέει μιλώντας για τα θέματα αυτά. Εγώ είμαι επικεφαλής λοιπόν της μονάδας που ασχολείται με το κλίμα, αλλά είμαι και επικεφαλής ε, με την εκπεριτροπή ε, ε, ομάδα του της Προεδρίας του Συμβουλίου ε, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και μάλιστα ε, κατά ε, όπως έγινε και προηγούμενες χρονιές όπως έγινε και στο Παρίσι που και ο εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου και η υπουργό ήταν γυναίκες και φέτος το ίδιο συμβαίνει είναι και η υπουργό και η εκπρόσωπος γυναίκες όσον αφορά την δράση για το κλίμα και νομίζω ότι ε, μπορεί κανείς ε, να πει με ασφάλεια ότι υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες οι οποίες ε, είναι πολύ σημαντικές και είναι αυτές ακριβώς οι προσωπικότητες οι οποίες άνοιξαν, διεύρυναν τη διάσκεψη των Παρισίων. Η συμφωνία του, του Παρισιού λοιπόν οπωσδήποτε όπως υπόθηκε ήδη πολλές φορές αποτελεί καμπή, αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο γιατί ε, δεν εστιάζει πλέον στον μετριασμό των αποτελεσμάτων όπως παλιότερα. Ε, η Συμφωνία των Παρισίων αναφέρεται ε, στην οικονομική υποστήριξη, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την μεταβίβαση γνώσεων. Στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης, η Συμφωνία των Παρισίων είναι δυναμική, είναι ειλικρινή κανείς έφερε ε, κοντά ε, όλους τους εμπλεκόμενους γιατί ε, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε μονάχα με, το καλό ας πούμε να συμφωνήσουν όλοι με στόχους σημαντικούς όπως ας πούμε το 1,5 λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κατάσταση, την αύξηση του επίπεδου των ωκεανών λοιπά Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στην διεθνή κοινότητα ε, να επανέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ε, να συζητάει, ε, να προσπαθεί να βρει λύσεις, να διορθώνει τις λύσεις που έχουν βρεθεί σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η Συμφωνία των Παρισίων είναι αποτέλεσμα διακυβερνητικής συνεργασίας και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν τα μέτρα, να ληφθούν ε, τα μέτρα και να τεθούν σε ισχύ ε, σε τοπικό επίπεδο μέσω συγκεκριμένων απτών μέτρων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που μιλάμε για στόχους του 2030 που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Έχουμε πολλές δεκαετίες εμπειρίας κλιματικής ε, πολιτικής που οπωσδήποτε έχουν ε, βοηθήσει ε, την μετατροπή της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία που σιγά σιγά ενδιαφέρεται για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και προσπαθεί να τις μειώσει. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα ε, ε, οι οικονομίες των χωρών του G20 ε, κινούν κατά 80% την οικονομία και την βιομηχανία και επομένως εκεί βρίσκεται το κλειδί και η απάντηση για τη μείωση των εκπομπών οι στόχοι, η η αναπτυξιακή ε, στόχοι ε, ε, μαζί για το 2050 μαζί με τη Συμφωνία των Παρισίων αποτελούν τα κύρια βήματα προς τα εμπρός και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να, να απελευθερωθούν οι συνέργειες μεταξύ των στοιχείων αυτών. Γνωρίζουμε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να δοθεί απάντηση και σε συγκεκριμένα συγκεκριμένα γεωπολιτικά προβλήματα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη όθηση, υπάρχει momentum ε, που μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή. Αλλαγή που είναι απαραίτητη έτσι ώστε να παραμείνουμε στην τροχιά που έχουμε χαράξει. Ε, ίσως να πω και δύο λόγια όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι η ενδυνάμωση των γυναικών, όπως και η δημοκρατία, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, η ισότητα των φύλων είναι στοιχεία απολύτως απαραίτητα. Ε, οι γυναίκες ε, είναι το πρωταρχικό στοιχείο της οικογένειας και κατά αυτή την έννοια ο ρόλος τους ε, είναι καταλητικός και ιδιαίτερα σημαντικός. Ένας από τους στόχους των κλιματικών συζητήσεων ε, είναι η πλήρης εμπλοκή των γυναικών ως προαπαιτούμενο για αποτελεσματική κλιματική ε, πολιτική. Ε, σαφώς αναφέρεται και ρητά στη Συμφωνία των Παρισίων ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους που έχουν παρόμοιες απόψεις. Επίσης ε, αναγνωρίζεται ε, η ανάγκη αυτού που είπε προηγουμένως ε, και η κυρία Ρόμπινσον, δηλαδή η ενδυνάμωση των γυναικών στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο στο προήμιο, αλλά και στο διατακτικό του κειμένου αναφέρονται αυτά τα στοιχεία, γιατί καμιά φορά το προήμιο είναι εκεί που μπαίνουν όλοι οι ευσεβείς πόθοι, αυτά τα στοιχεία αναφέρονται και στο διατακτικό. Ε, συγκεκριμένα μιλώντας, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργά συμμετέχει ε, στην διαμόρφωση προγράμματος συμμετοχής των γυναικών και ενδυνάμωσης των γυναικών και τα ξέρω από πρώτο χέρι γιατί έχω συμμετάσχει σε όλες τις διαπραγματεύσεις αλλά ε, επίσης είμαστε και από τους φορείς που χρηματοδοτούν ε, την, ε, τις διαδικασίες ενδυνάμωσης των γυναικών. Με προσοχή ακούω οτιδήποτε προέρχεται και από τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά την ισότητα των γυναικών και αυτά που άκουσα με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω όλα αυτά τα μέτρα Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες και έχει ολοκληρωμένα και διευρυμένα προγράμματα με τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κατανοούμε ε, πόσο σημαντικό είναι ε, να μελετήσουμε τα, τα στοιχεία αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αξιολογεί, κάνει μια εργασία αξιολόγησης της προσαρμογής και της διαδικασίας αξιολόγησης έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να προσαρμόσουμε την στρατηγική μας, διότι η στρατηγική προσαρμογή θα πρέπει με τη σειρά της να προσαρμόζεται ε, σε τακτά διαστήματα βάσει των πιλωτικών δράσεων. Όσον αφορά την συνεργασία, ε, να πω ότι συνεργαζόμαστε στενά με την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ε, όχι μόνο για θέματα κλιματικής αλλαγής, αλλά και για θέματα συμπερίληψης και για θέματα κοινωνικής ισότητας, ισότητας των γυναικών κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τμήματα του γενικότερου δόγματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τελειώσω λέγοντας ε, ότι εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ σοβαρά ε, με την κλιματική δικαιοσύνη και την ισότητα των γυναικών. Ε, συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους μας έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να αποτελούν τμήμα όλων των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους, με όλες τις ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τις αρχές αυτές έτσι ώστε να ε, διαβουλεύετε μαζί τους, να ακούει την άποψή τους για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κυρία Μπάρντρα. Η επόμενη καλεσμένη μας είναι η Στεφάνια Δελζότη, υπεύθυνη προγράμματος στη μη κυβερνητική οργάνωση «Ο κόσμος από τη σκοπιά των γυναικών». Um, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καλέσατε την κυβερνητική οργάνωσή μας ε, σε αυτή την ακρόαση και να εκφράσω την τιμή που νιώθω για την παρουσία μου εδώ. Καταρχήν η μη κυβερνητική αυτή οργάνωση, ο κόσμος από τη Σκοπιά των Γυναικών, είναι βελγική μη κυβερνητική οργάνωση που ε, εστιάζεται στις γυναίκες ε, και την ανάπτυξή τους υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων και εμπλεκόμαστε σε κοινωνικά κινήματα την τελευταία 20 ετία. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και την αλληλεγγύη και στο Βορρά και στο Παγκόσμιο Νότο σε συνεργασία με πολλές ε, οργανώσεις στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Και μάλιστα εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ανταλλαγή απόψεων με, με, μεταξύ ισοτήμων για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις, κάτι που χρειαζόμαστε και στην περίπτωσή μας. Είχα ετοιμάσει μία παρουσίαση με PowerPoint, αλλά έχει πλέον ξεπεραστεί μετά τις τελευταίες ομιλίες. Γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε μερικά κέρια σημεία για να τροφοδοτήσω τη συζήτηση. Καταρχήν να κάνουμε κάποιες προκαταρκτικές αναλύσεις. Ε, βλέπουμε ότι εξακολουθούν να, να παρατηρούνται διαρθρωτικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βέβαια, οι γυναίκες δεν είναι μια ομοιογενής ομοιόμορφη ομάδα και το γεγονός ότι είναι κανείς κάποια γυναίκα αποτελεί βασικό λόγο για να υφίσταται διακρίσεις στον κόσμο. Έχουν ε, συνταχθεί πολλές μελέτες και έχουν γίνει πολλές έρευνες που καταδεικνύουν τον αντίκτυπο που έχουν οι κλιματικές αλλαγές ε, στις γυναίκες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτές τις αλλαγές και βλέπουμε τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, κυρίως γιατί σε πολλές χώρες ε, αυτές φροντίζουν για το νοικοκυριό και για τον βιοπορισμό της οικογένειας, συμμετέχουν στην παραγωγή τροφίμων και φυσικά επηρεάζονται από την κατάσταση μεταξύ των δύο φύλων. Άλλωστε, το θέμα της ισότητας των φύλων αφορά ένα κοινωνικό πλαίσιο, το ρόλο και τις κωδικοποιημένες σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και αφορά και το σχετισμό δυνάμεων, τη σχέση ισχύω, έχει κάποια, κάποια συνέπειες στην ιεραρχία και φυσικά επιδέχεται αλλαγές ε, και στο χώρο και στο χρόνο. Αν υιοθετήσουμε λοιπόν μία προσέγγιση από τη σκοπιά του φύλου, μπορούμε να περιλάβουμε εκεί και την πρόθεση τη συμμετοχή των γυναικών, που έχει κέρια σημασία, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποια στερεότυπα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε και τις διαρθρωτικές ανισότητες. Και μια και οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες από άποψη φύλου, θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και στις διαπραγματεύσεις μας για τις κλιματικές αλλαγές και τις συναφείς πολιτικές. Επίσης, ε, η εφαρμογή και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθεί να συνιστά μεγάλη πρόκληση. Δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων ε, σχετίζεται με μακροπρόθεσμες αλλαγές, αλλαγή νοοτροπίας, ε, συμπεριφοράς, στάσεις οι μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς πολιτική βούληση, χωρίς διαφάνεια, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο και φυσικά επαρκή προϋπολογισμό. Ε, ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο και ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα από μια κυβερνητική οργάνωση με την οποία συνεργαζόμαστε στη, Βολιβία, τη ΡΕΜΤΕ. πρόκειται για ένα δίκτυο ε, με θέμα το πώς μπορούν οι γυναίκες να αλλάξουν την οικονομία και συμμετείχαμε σε τριετή προγράμματα προωθώντας τις παραδοσιακές γνώσεις των γυναικών συμπεριλαμβάνοντας και τις δικές τους ε, συστάσεις και προτάσεις σε δημόσιες πολιτικές όπως αυτή για τις κλιματικές αλλαγές. Ε, το πρώτο μας εγχείρημα αφορούσε κάποια έρευνα ε, συνεργατικής δράσης με πανεπιστημιακούς, αλλά και τοπικές οργανώσεις και τοπικές κοινότητες. Και στη δική μας κυβερνητική οργάνωση, αλλά και σε πολλές άλλες οργανώσεις ε, ε, πιστεύουμε, όπως και οι ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών, θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινούμε εκ του μηδενός και μία από τη βάση προς τα πάνω, συνδέοντας τους ακαδημαϊκούς κύκλους, τους πανεπιστημιακούς με τις τοπικές κοινότητες, ώστε να αποκομίσουν εντυπώσεις για την πραγματικότητα και το πώς τη βιώνουν αυτοί καθημερινά οι γυναίκες. Ήταν ε, σημαντικές ριζικές ε, οι αλλαγές στη ζωή των γυναικών, μεγαλύτερη έκθεσή τους σε θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Επίσης, ε, η δυσκολία στην προβλεψιμότητα των βροχών δυσκόλεψε και την παραγωγή τροφίμων. Είναι ε, δύσκολη πρόσβασή τους στο νερό, ε, ο φόρτος εργασίας τους αυξάνεται και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα κυριαρχίας ε, παραγωγής τροφίμων, ώστε με αποτέλεσμα να έχουν ελάχιστο χρόνο ελεύθερο ή να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, σε συναντήσεις. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η μετανάστευση οι άντρες πήγαιναν προς τις μεγάλες πόλεις να εργαστούν, είτε και οι γυναίκες μερικές φορές ε, έπρεπε να μετικήσουν. Και μάλιστα όταν ασχολούνται με τα, όταν ασχολούνται με τα οικιακά ήταν πολύ πιο εκτεθειμένες στην ενδοικογενειακή βία και στα συναφή ζητήματα. Σε περίπτωση που οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι για απασχόληση. Επίσης, ε, ήταν σημαντικό να δείξουμε ότι οι γυναίκε ήδη δρούν πολύ συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν τι παραδοσιακέ του γνώσει για τη γη και βρίσκουν εναλλακτικέ λύσει για να μετριάσουν μερικά από τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών. Για παράδειγμα, έχουμε άμυψη σπορά, βιολογικά λιπάσματα, διαχείριση αποβλήτων και ούτω καθεξής. Ε, δεν θα επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειες. Το σχέδιό μας ε, προσπάθησε να στηρίξει και τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις ε, και καλύτερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προτάσεις ε, σε πολιτικές πρόληψης και μετριασμού και συμμετοχή σε έλλειψη αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Βέβαια, είχαμε και ένα προηγούμενο σχέδιο με το ίδιο περιεχόμενο, επίση του Διάρκεια, που συνέβαλε πολύ στη χειραφέτηση των γυναικών, στην ενίσχυσή τους και άνοιξε το δρόμο και για το δικό μας σχέδιο, γιατί έδειξε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των γυναικών στην εξασφάλιση της ε, αυτάρκειας, της κυριαρχίας και της παραγωγής των τροφίμων. Επίσης ασχοληθήκαμε με την με τις τεχνικές δυνατότητες για την δημιουργία ικανοτήτων και είχαμε ανταλλαγές απόψε με αντίστοιχες γυναικείες οργανώσεις της περιοχής. Και φυσικά οι γυναίκες δεν διεκδικούσαν μόνο τα δικά τους δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά επέμειναν και στα δικαιώματα της μητέρας γης, του πλανήτη μας. Εξού και η σημασία του να συμπεριλάβουμε την έννοια της ευζοίας, του ευζήν, Bien στις ε, διαπραγματεύσεις για το κλίμα και το περιβάλλον. Το δικαίωμα δηλαδή να ζει κανείς μία αξιοπρεπή ζωή, μία αξιόλογη ζωή. Και φυσικά εδώ χρειάζεται μία πιο μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τις τοπικές αυτές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και από αυτή την άποψη η Βολιβία μπήκε στον κατάλογο των χωρών μέσου εισοδήματος παρόλο που δυστυχώς ακόμη και στις πλουσιότερες χώρες οι πλέον ευάλωτες ομάδες εξακολουθούν να παραμένουν ευπαθείς και ευάλωτες. Και αυτή η διάκριση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί το ΑΕΠ δεν είναι κατάλληλο μέσο υπολογισμού ή αξιόπιστος δείκτης για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό λοιπόν ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασία. Είχα προετοιμάσει και κάτι για τα δικαιώματα των γυναικών και τι κλιματικέ αλλαγέ, μια και όμω αυτό το θέμα ήδη καλύφθηκε από τι προλαλήσει σα. Θα το περάσω. Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε το θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη για το κλίμα, γιατί συμβάδισαν ε, εκ παραλίλου, συμβάδισαν για μεγάλο διάστημα Πάντω Ρίο, από το Ρίο το 1992 έγινε μια, ε, ε, ένα συνδυασμό τους, οπότε ε, με την διακήρυξη του Ρίο έχουμε το πρώτο δημόσιο, ε, το πρώτο διεθνές εργαλείο που αναγνωρίζει τη σημασία της ανάμειξης και της εμπλοκής των γυναικών. Και στην COP22 ε, πέρυσι το φθινόπωρο στο Μαρακές, το ενδιαφέρον ήταν ότι Έχουμε πλέον κατοχύρωση της αρχής της, συνε... της συνοχής μεταξύ των διεθνών ε, πολιτικών και των ε, παγκοσμίων ε, μέσων και διακηρύξεων όπως ε, του Διεθνούς Σχεδίου Εργασίας της Αντισαμπέμπα και άλλων όπως η διακήρυξη του Πεκίνου και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία μιας ε, διαδήλωσης ε, γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι οι, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το περιβάλλον και αυτές για την ισότητα φύλου θα πρέπει να ε, συσπηρωθούν, να συνεργαστούν και να ενώσουν τις δράσεις τους. Κάτι που συμβαίνει όλο και περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, συνεργαζόμαστε με ε, εταίρους, άλλες οργανώσεις μη κυβερνητικές, γυναίκες ή γυναικείες οργανώσεις, εκτενής ο κατάλογος, δεν πρόκειται να διαβάσω όλες τις συστάσεις. Πάντως αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διαπραγματεύση θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, από το τοπικό έως το παγκόσμιο. Υπάρχει και το θέμα της μελέτης επιπτώσεων από τη σκοπιά του φύλου και επίσης το θέμα της αντιμετώπισης των διαρθρωτικών ανισοτήτων, κάτι που όπως είπα υπερβαίνει την συμπερίληψη κάποιων κριτηρίων ισότητας φύλων. Επίσης, υπάρχει το θέμα των ε, ε, σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, της πρόσβασης ε, των γυναικών στη γη και στον έλεγχο της γης και την πρόσβαση στους σπόρους και υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης, που είναι ένα άλλο από τα θέματα που θα αναλύσω στη συνέχεια. Ήθελα εδώ να σας δείξω αυτή τη μάνταλα, δυστυχώς είναι στα γαλλικά. Είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνεργασίας ε, με ε, οργανώσεις ε, εταίρους που δείχνει ότι η χειραφέτηση δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα, γιατί συνήθω αυτό λαμβάνεται υπόψη όταν μιλούμε για ενίσχυση ή χειραφέτηση των γυναικών, μόνο το οικονομικό σκέλο, αλλά εδώ θέλουμε να δείξουμε ότι τοπικές γυναικείες οργανώσεις ε, αντιμετωπίζουν τη χειραφέτηση σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο και φυσικά ε, είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο, γιατί όταν λέμε για παρόν εννοούμε ε, υπεροχή, ενώ όταν μιλούμε για παρόφ μιλούμε για έλεγχο της γνώσης των πόρων, επίσης μιλούμε για ε, δέσμευση, αλληλεγγύη και το power within που προϋποθέτει η αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να κάνει κανείς τις προσωπικές του επιλογές ελεύθερα. Οπότε βλέπετε πόσο πολυσύνθετο είναι το θέμα της χειραφέτησης και σίγουρα δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση χειραφέτησης των γυναικών. Ποια είναι τώρα τα κέρια ζητήματα που θα κληθούμε να λύσουμε, ποιες οι βασικές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα της, των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στις ε, περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να διαχωρίζεται από το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το, της αποτελεσματικότητας. Η συμμετοχή των γυναικών έχει προταθεί κυρίως ως κάτι αποτελεσματικό, ενώ είδαμε στο Μαρακές ότι αλλάξαμε κάπως το πρίσμα και το συνδέσαμε με την προσέγγιση που εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, οι γυναίκες ήδη δραστηριοποιούνται, ήδη είναι ενεργές και ε, συμμετέχουν επαρκώς, θα πρέπει όμως να ε, είναι παρούσες ε, και να ακούγεται η φωνή τους και στις διαπραγματεύσεις. Ο, επίσης, ο ο τρόπος σκέψης ε, και οικονομικής ανάπτυξης είναι προβληματικός. Τώρα, ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στη μη αμοιβόμενη γυναική εργασία ή στην ιδέα των ανεξάντλητων φυσικών πόρων είναι ένα βιώσιμο μοντέλο ή μήπως όχι. Επίσης, κάποιες συγγραφείς κάνουν παραλληλισμό μεταξύ της ε, αντιμετώπισης ε, των γυναικών ως αγαθών, ως εμπορευμάτων και της αντίστοιχης αντίληψης για τη φύση. Πόσο δηλαδή και η φύση και οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο ή ως εμπόρευμα. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας ως απόρρια κάποιων φυσικών καταστροφών, θεομηνιών ή κλιματικών αλλαγών. Επίσης υπάρχει μεγάλη βία εις βάρος των γυναικών σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Δεν είναι όλα τα θέματα αυτά ασύνδετα. θα πρέπει λοιπόν να δούμε την αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, εδώ έχουμε και βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, τη υφαρπαγή των γεών. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν δεόντως. Επίσης, κάτι που είπε η κυρία Ρόμπινσον, είναι σημαντικό να ακούμε ένα τον άλλον, να αφογκραζόμαστε ε, και να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Και αυτό γίνεται και διακλαδικά αλλά και σε ε, πολλά επίπεδα. Επίσης, η κρίση δίνει και ευκαιρίες. Και με τις αναδυόμενες απειλές και τη δίνει μερικές φορές πραγματικότητα, θα πρέπει να βρούμε την ευκαιρία να εργαστούμε για ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή να θέσουμε στόχους και να προβλέψουμε και επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Αυτά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εσάς. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, τελευταία ομιλητήρια, την κυρία Στάφανσον. Dear all, dear all women, dear all men. Από το Αρκτικό Συμβούλιο, Σάμι. Κυρία Στάφανσον. Άλλη ε, δηλώνουν, ε, υπάρχουν κάποιοι που δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε κάποιο φύλλο ή ανήκουν σε κάποια από τα άλλα φύλλα, όχι τα δύο. Εγώ καλωσορίζω τους πάντες και έχω έρθει εδώ να σας πω τη δική μου ιστορία. Λέγομαι Γιάννη, γεννήθηκα ε, σε μια οικογένεια που ε, εκτρέφει ταράνδους και εξακολουθώ να ζω εκεί όταν ε, είναι ήρεμοι τάρανδοι και τους προσέχουμε, είναι πολύ χαρούμενοι και είμαστε και εμείς χαρούμενοι και ο ίδιος κανόνας ε, ισχύει. Εργαζόμαστε και στο Συμβούλιο το Αρκτικό ε, για τους ίδιους λόγους με το λαό Σάμι που είναι οι μόνοι αυτόχθονες στην Ευρώπη. Ζούμε στη βόρεια Σκανδιναβική Ήπειρο και στη βορειοανατολική Ρωσία. Όπως όλοι οι αυτόχθον πληθυσμοί, και εμείς έχουμε στενές σχέσεις με τη φύση, με τη γη και το περιβάλλον. Και έχουμε αναπτύξει εργαλεία για να καταλαβαίνουμε, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τη φύση και να επικοινωνούμε μαζί της. Έχουμε αναπτύξει εργαλεία για να ακούμε τα μοτίβα της, ε, και να τα, της φύσης και να τα παρατηρούμε. Όμως εδώ και 25 χρόνια σταμάτησε να μας δίνει αυτά τα μοτίβα η φύση και είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρουμε ε, τι συμβαίνει. Είναι σαν να έχει αγχωθεί κατά κάποιο τρόπο. Άλλοτε δεν έχουμε κάποιες εποχές που είχαμε, ενώ υπάρχουν ε, άλλες εποχές που δεν είχαμε. Είναι σαν να έχουμε 8 εποχές. Όλα αυτά επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι όμως απειλή. Είναι κάτι που είναι εδώ. Είναι ένα σοβαρό θέμα βέβαια. Για εμάς κεντρική σημασία έχει ο καιρός. Το συζητάμε κάθε βράδυ στο τραπέζι. Και κάθε μέρα προσπαθούμε να προβλέψουμε τον καιρό. Γιατί από τον καιρό εξαρτάται η ζωή μας. Και η ζωή των ταράντων που εκτρέφουμε. Θέλουμε να δούμε ε, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για, τις, για τα καιρικά φαινόμενα, όπως και εσείς βέβαια. Ανήκω στη γενιά της αλλαγής του κλίματος και έχω ακούσει τους πιο μεγάλους ε, για την αλλαγή του κλίματος και πραγματικά είναι ανησυχητικά όλα αυτά, δεν φαίνονται καθόλου αισιόδοξα, όμως αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να τις κάνουμε και τις δράσεις τις απαιτούμε, θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να λάβουμε σκληρές αποφάσεις για πολιτικές που αφορούν την καθημερινότητά μας. Χρειάζεται επίσης μια συστημική αλλαγή και μια αλλαγή ζωής για όλους. Ίσως πολλοί από εσά θα σκέφτεστε πώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή μας συνέχεια έλεγε του κλίματος. Εγώ με τους θάνατους για παράδειγμα. Ανάλογα με το πώς είναι ο καιρός, θα πρέπει να τους βρω ε, τόπο να βοσκήσουν, να πρέπει να τους μεταφέρω σε ασφαλές σημείο και αλλάζουν ε, καιρικές συνθήκες συνέχεια. Μέσα σε 12 ώρες μπορεί να αλλάξουν ε, οι θερμοκρασίες 35 βαθμούς ε, ε, έχουμε περιοχές τιμών, μπορεί να έχουμε ε, πάγο, μπορεί να έχουμε αντίστοιχα να σπάει ο πάγος ε, λόγω της απόταμης ανώδης θερμοκρασίας και έτσι οι τάρανδοι δεν μπορούν να βοσκήσουν εκεί που συνήθιζαν να βοσκήσουν. Θα πρέπει να βρούμε νέους βοσκοτόπους. Επίσης, η βροχή είναι κάτι που υποτίθεται δεν θα έπρεπε να συμβαίνει το χειμώνα, αλλά συμβαίνει. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μόνο πάγο. Επίση, πρέπει να πω ότι οι τάραντι που μπορούν να μυρίζουν ε, την τροφή του κάτω από τον πάγο δεν μπορούν πλέον να σμιστούν ε, την ε, μετάπαυση πάνω στην κρούστα του, του πάγου αυτή την τροφή, τη, τη βοσκή. Επίσης πρέπει να σας πω ότι όταν ε, βρέχει ενώ κάνει ακόμα πάρα πολύ κρύο, αυτό είναι φανατική καταδίκη για τους ε, νεογέννητους ταράδους. Ε, και το είδα και στα μάτια της αδερφής μου, πραγματικά τον πόνο που ένιωθε, γιατί ήξερε ότι αυτά τα νεογέννητα δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Υπάρχει επίσης άλλο πρόβλημα. Στις λίμνες δεν είναι σταθερός ο πάγος. Αλλάζουν ε, οι συνθήκες και στα ποτάμια και στις θάλασσες. Ε, μπορούσαμε να διασχίσουμε τις παγωμένες λίμνες, τα παγωμένα ποτάμια. Τώρα δεν είναι ασφαλές αυτό και για τους θανάδους. 300 τάρανδοι ε, πρόσφατα κάποια χρονιά έχασαν τη ζωή τους πέφτοντα στα παγωμένα νερά, επειδή έσπασε ο πάγο και εμεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρά να του βλέπουμε να πεθαίνουν. Έχουμε χάσει και πολλούς ε, ανθρώπους λόγω της αλλαγής του κλίματος ε, και λόγω του τρόπου κατανάλωσης και τρόπου ζωής των άλλων. Εμείς πληρώνουμε. Πληρώνουμε το δικό μας το αίμα. Εγώ ε, πλήρωσα με την οικογένειά μου και ίσως και στο μέλλον θα συμβεί κάτι αντίστοιχο αν δεν αλλάξει το, ο τρόπος μας, αν δεν έχουμε μια συστημική αλλαγή. Θα πρέπει να αλλάξουμε μοτίβα, να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αλλάξουμε τρόπο ζωής με τις ποιες ενέργειες, με την πράσινη ενέργεια βέβαια, ε, πρέπει να ξέρετε ότι και ευθύνη είναι μεγάλη, διότι στον πλανήτη σήμερα πολλοί αυτόχθονοι πληθυσμοί βλέπουν τα δικαιώματά τους να ε, παραβιάζονται, να καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω ακριβώς της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Και εγώ είμαι υπέρ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Φυσικά γιατί χρειαζόμαστε την πράσινη ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καταπατούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων μεταξύ των ηγετών των αυτοκθόνων είναι πολλέ γυναίκες και πολλοί νέοι. Και πραγματικά πολλές φορές παρενοχλούνται, απάγονται, για να μην πω δολοφονούνται, επειδή ε, υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους, ε, τη γη τους ε, και τη φύση ουσιαστικά. Σήμερα στη Σουηδία υπάρχουν πολλές κοινότητες οι οποίες αγωνίζονται κατά τεράστιων λοιπόν πάρκων που υποτίθεται ότι θα ε, ανεγερθούν ακριβώς εκεί που ζουν οι τάρανδοι, άρα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ε, τάρανδων, που δεν πρόκειται να πλησιάσουν σαν γεννήτριες. Ε, ε, και αυτοί οι οποίοι θα καταναλώνουν την ενέργεια αυτή ζουν πάρα πολύ μακριά από αυτά τα εδάφη και στη δεκαετία του 50 αλλά και το 19ο αιώνα όταν είχαμε μια νέα εξέλιξη με εργοστάσια που φύγαμε, χάσαν τη, βοσκοτόπια του Σιτάρανδη και πληρώσαμε βαρύ τίμημα, ε, βαρύ φόρο. Και επειδή ζητάμε την αηφόρα να δείξει την ενέργεια αυτή, ποιος την πληρώνει όμως. Και ποιο, ποιο είναι το τίμημα των καταναλωτικών αναγκών σας. Εγώ την ξέρω την τιμή, το ξέρω το τίμημα. Όταν έχουμε λοιπόν αυτή τη μετάβαση, ακριβώ τότε είναι που χρειαζόμαστε και την κλιματική δικαιοσύνη. Πρέπει να έχουμε αυτή τη βιωσιμότητα, αυτή την αηφορία. Δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμε εξορυκτικές βιομηχανίε ή πράσινη εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι κάτι που πρέπει να το υπερβούμε. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε, να το δούμε αλλιώ το πράγμα. Και γι' αυτό ήρθα εδώ για να σας τα πω αυτά σήμερα, που είναι η πρώτη ακρόαση για θέματα κλιματικής δικαιοσύνης και σας χειροκροτώ πραγματικά. But what took Γιατί αργήσατε όμως τόσο πολύ. Τι κάνατε τόσο καιρό. Και έχω και μια πρόκληση να σας απευθύνω. Σε ό,τι αφορά την κλιματική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι κάτι που μόνο αποδίδεται σε αυτούς που μπορούν να επικοινωνούν στη δική σας γλώσσα. Με ανθρώπινη μορφή. ή και άλλοι δικαιούνται ακριβώς την απονομή δικαιοσύνης. Δεν έχουν άλλοι δικαιώματα. Μόνο τα δικά σας παιδιά. Τα δικά σας παιδιά, τα νεογέννητα έχουν δικαιώματα. Τα ζώα που δεν μπορούν να μιλήσουν ή να επικοινωνήσουν στη δική σας γλώσσα ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όπως εμείς έχουν δικαιώματα. Τα φυτά έχουν δικαιώματα. Τα ποτάμια έχουν δικαιώματα. Η γη έχει δικαίωμα. Με αυτή την αντίληψη περί κλιματικής δικαιοσύνης, για μένα τουλάχιστον, όλα τα όντα περιλαμβάνονται. Συγκεκριμένα στη Νέα Ζηλανδία ε, απέκτησε νομική προσωπικότητα ένα ποτάμι. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο καθεστώς των δικαιωμάτων της μητέρας γης, τα δικαιώματα των ποταμιών, της αγέννητης γενιάς. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 25 λεπτά για παρεμβάσεις ε, από, τους, ε, το ακροατήριο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Και θα δούμε αν έχουμε μετά χρόνο και για δεύτερο γύρο. Μαρία, ευχαριστώ Μέρη. Θα μιλήσω γαλλικά να βάλετε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, λέει η κυρία Ρενά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, μαρτυρίες ε, που ακούσαμε από σας σήμερα. Είμαι υπερήφανη που συμμετέχω σήμερα σε αυτήν τη συζήτηση στην Επιτροπή Γυναικών, Επιτροπή που συχνά θίγει θέματα τα οποία δεν θίγονται σε άλλες ε, επιτροπές ε, με την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει όπως είπατε και εσείς ότι θα αλλάξουν τα πράγματα έστω και αν δεν είναι πάντα ευνοϊκές οι καταστάσεις ε, η ελπίδα υπάρχει και η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών δεσμεύεται σε αυτές τις διαδικασίες. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που ακούστηκαν όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο πάντως να δούμε το πρόβλημα του μοντέλου. Είναι κρίμα που η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει φύγει. Ε, βέβαια πιστεύω ότι κάποιος άλλος εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι εδώ. Αλλά παρόλα αυτά ε, πρέπει να τονίσουμε το θέμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην ΔΕΒ, στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΒ, τη Γενική Διεύθυνση ε, ΔΕΦΚΟ, τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, ε, που διαπραγματεύεται την αλλαγή του μοντέλου. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχω την τύχη να συμμετέχω και σε μια άλλη επιτροπή. Είναι η Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου. Και παραδόξως τη στιγμή που το διεθνές εμπόριο είναι ακριβώς αυτό το οποίο ε, εν τέλει ενισχύει το εντατικό μοντέλο το οποίο ε, ζούμε, ενισχύει την παραγωγή ε, που ενισχύεται ούτως ή άλλως από την επιταχυμένη ε, παγκοσμιοποίηση. Εγώ δεν είμαι κατά της παγκοσμιοποίησης, αλλά αυτή η επιταχυμένη ε, παγκοσμιοποίηση ε, οδηγεί σε μοντέλα τα οποία τελικά και στην Ευρώπη και αλλού θα ενισχύσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Το Κοινοβούλιο μάλιστα είδαμε ότι ε, ε, ε, εν τέλει έδωσε και πράσινο φως για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου. Επομένως, από τη μία μεριά υπογράφουμε την COP21 και από την άλλη συμφωνούμε, ε, υπογράφουμε ε, συμφωνίες με τον Καναδά ε, που είναι χώρα η οποία ακριβώς επιτρέπει τέτοιες εκμεταλλεύσεις και επομένως δεν σέβεται τις αρχές. Έχουμε επίσης συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Γκάνα. Είχα την τύχη να πάω εκεί με την συνάδελφο Χαουτάλα την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε την καταστροφή που έχει προκαλέσει η ε, Συμφωνία Ελεύθερων ε, Ανταλλαγών που έχει προκαλέσει κατάρρευση ε, του αγροτικού συστήματος και που ε, δημιουργεί πρόβλημα ε, και στις μικρές καλλιέργειες ε, τις οποίες παραδοσιακά είχαν οι γυναίκες. Δηλαδή από τη μία κατακριμνίζεται η οικονομία, φτωχαίνει η χώρα, φτωχαίνουν όμως και οι γυναίκες οι οποίες ήταν αυτές οι οποίες έφερναν το ψωμί στις οικογένειές τους. Επομένως έχουμε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κάνα που τελικά κανένα καλό δεν φέρνει. Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή Γυναικών πολύ καλά κάνουμε και συζητάμε για τέτοια θέματα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες επιτροπές όπως είναι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου στο Κοινοβούλιο πολλή δουλειά πρέπει να γίνει. Έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια σχιζοφρενική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια πλειοψηφία που στην Επιτροπή Γυναικών ε, ε, θα αποφανθεί ότι ναι πρέπει να δουλέψουμε υπέρ των γυναικών κτλ. και η ίδια πλειοψηφία όταν βρίσκεται στην Ολομέλεια ή σε μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή ε, θα ε, ε, συμφωνήσει, θα δώσει πράσινο φως σε καταστροφικές συμφωνίες. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς, εμείς που είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον εαυτό μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλουμε ε, πιο ε, θετική ε, σκέψη και πιο συνεκτική πράξη. Πολύ συχνά η Κομισιόν ενεργεί μόνη της. Να πω και κάτι τελευταίο όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών. Δουλεύουμε πολύ, συνεργαζόμαστε πολύ με την κοινωνία των πολιτών και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Αλλά αλλά νομίζω ότι τώρα ε, ε, ε, βάζουμε πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους της κοινωνίας των πολιτών. Αν δούμε την οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν αντέχει πια η κοινωνία των πολιτών. Εμείς ερχόμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους της σε χώρες του Νότου. Αυτή η κοινωνία δεν αντέχει των πολιτών, δεν αντέχει πια απέναντι στα λόμπις ε, γιατί εν τέλει πληρώνουν πολύ ακριβά την ελευθερία ε, που πετυχαίνουν για να κάνουν αυτά που θέλουν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μην υπερφορτώνουμε την κοινωνία των πολιτών, γιατί συχνά την παίρνουμε σαν άλοθη για να μην δουλέψουμε εμείς αρκετά σωστά και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τον κόδωνα κινδύνου που κρούει αυτή η κοινωνία των πολιτών και να αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες μας σχετικά με το μοντέλο το οποίο επιβάλλουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χάιντε Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορικές και εντυπωσιακέ παρεμβάσεις σας. Πριν από δύο χρόνια Είχα μια σοκαριστική αλλά και ε, ενδιαφέρουσα εμπειρία μαζί με το Carbon Watch αλλά και σε, με άλλες ε, οργανώσεις. Είχαμε μια συνάντηση εδώ ε, και ήρθαμε σε επαφή με θύματα μιας κατάστασης αντίστοιχης με αυτήν που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Στάφανσον. Ε, δηλαδή κάποια προγράμματα τα οποία άλλαξαν ριζικά άρδιν τις ζωές των ανθρώπων αυτών. Όμως αυτό το πρόγραμμα είχε τη σφραγίδα του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Κάποιοι συνάδελφοι μαζί με μένα, δύο-τρεις είμαστε, ε, αμφισβήτησαν τις διαδικασίες ε, του καθαρού μηχανισμού ε, των Ηνωμένων Εθνών. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω αν άλλαξε κάτι. Ίσως ε, θα τα λάβει υπόψη της ε, η συνάδελφος Λίνα Έγκστρομ στην επόμενη έκθεσή της. Θέλω να πω ότι ακόμα και διεθνείς οργανισμοί κάνουν, παίρνουν αποφάσεις οι οποίες τελικά ε, κάνουν ακόμα δυσχερέστερη την ε, ήδη δυσχερή και δυσμενή θέση των γυναικών. Επομένως ε, είναι πάρα πολύ καλό που ακούμε ότι δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι στο Αρκτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα τουλάχιστον στην Αρκτική. Μέρι Ρόμπινσον, ξέρουμε ότι έχεις εμπλεκεί σε διεθνέ επίπεδο στα θέματα της κλιματικής αλλαγή. πιστεύει ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία, υπάρχουν δυνατότητες πραγματικά να λύσουμε προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Χάουντι. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στα καταληκτικά σχόλια. Άλλο κανεί. Πετήρ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις καλεσμένες μας για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν. Φυσικά, όλοι θα πρέπει με τη δέουσα σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, γιατί μπορούν να αποσταθεροποιήσουν και τον κόσμο ολόκληρο και το επιμέρους κράτη, αν δεν κάνουμε όλοι ότι μπορούμε όλα τα κράτη προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και σίγουρα οι γυναίκες και οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες. Αν δεν εξασφαλίσουμε ε, χρηματοδοτική υποστήριξη, επιστημονική έρευνα και μια ε, νομική ε, διάρθρωση διαχείρισης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, τότε θα αναχαιτήσουμε την ανάπτυξη και θα δημιουργηθούν συγκρούσεις για την πρόσβαση στο νερό, τα τρόφιμα και τις γεωργικές εκτάσεις. Θα αυξηθεί η φτώχεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε παγκόσμια αλληλεγγύη και κοινέ προσπάθειες για να μειώσουμε τους κινδύνους από τις κλιματικές αλλαγές που μας περιμένουν. Γιατί οι κλιματικές αλλαγές είναι κάτι που ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά και καμία χώρα, κανένας λαός από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, να μετριάσει τις κλιματικές αλλαγές. Χρειάζεται συνεργασία και κοινή δράση και επίσης συγκεκριμένα μέτρα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την εφαρμογή τους. Η ΔΕΜΗ θα έχουμε μαζικές μεταναστευτικές ροές γιατί οι κλιματικές αλλαγές περιορίζουν τους φυσικούς πόρους και απειλούν την ίδια την παραγωγή των τροφίμων θα έχουμε καύσονες, επιδημίες, ε, λοιμώδεις ε, νόσους ε, που θα απειλήσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Γι' αυτό είχαμε πρόσφατα πόσο οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και ζωή. Επίσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, επιστημονικές έρευνες που έγιναν στη Μασαχουσέτη και που προειδοποιούν κρόν τον να του κινδύνου για το πώς οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν και το δημογραφικό τοπίο. Για παράδειγμα, έγιναν έρευνες ε, για τις Ηνωμένε Πολιτείε που λένε ότι μέσω του 1991 και το 2000 ε, κάθε ημέρα με καύσον είχαμε 1165 καθυστερήσεις σε γεννήσεις. Και αυτό θα δημιουργήσει συγκεκριμένα προβλήματα και γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, σε θέματα όχι μόνο στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Δεν είναι αυτό ο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τι ειδικές ανάγκε των γυναικών και τα προβλήματά του ή τι μελλοντικέ απειλέ. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα και να δούμε πώ θα βοηθήσουμε αυτού που είναι πιο ευάλωτοι και πιο εκτεθειμένοι στι απειλέ. Ένα από τα μέτρα θα ήταν ίσω καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Μάλιστα, επειδή είμαι συνσηγήτρια για το θέμα αυτό, θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των γυναικών για την εξασφάλιση αυτή της ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες ε, τις συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Δεν υπάρχει άλλη ομιλήτρια ή ομιλητή στον κατάλογό μας. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στις καλεσμένες μας για να ολοκληρώσουν. Δύο-τρία λεπτά στην καθεμία παρακαλώ, γιατί στις 5.30 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και στο τέλος θα δώσω το λόγο στη Μέρι Ρόμπινσον για να κάνει μια σύνοψη ανακεφαλαίωση και μετά στην εισηγήτρια για πολύ σύντομα καταληκτικά σχόλια θα ακούσουμε τις καλεσμένες μας με τη σειρά που μίλησαν και προηγουμένως. Πρώτα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σχολιάσω κάτι που είπατε για την πολιτική και ε, εγώ ε, αντιμετωπίζω αυτά τα θέματα υπό τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ για την αναπτυξιακή συνεργασία. και το θέμα τη συνοχής των πολιτικών είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη. Αλλά πολλέ τρίτε χώρε προσδιορίζουν ίδια στο αναπτυξιακό τους μοντέλο και ε, εφόσον επιδιώκουν εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσει με άλλες ομάδες έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Τώρα, το ζητούμενο για μας είναι να εξασφαλίσουμε μία επαρκή διαδικασία διαβούλευσης και στις χώρες αυτές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ομάδων που ε, είναι σκόπιμο να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις. Και από την Αναπτυξιακή Σκοπιά εξετάζουμε το θέμα της συνοχή των πολιτικών ε, στις διάφορες δραστηριότητες μας. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω για το θέμα των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών δεν είμαι αρμόδια γι' αυτό. Και επανέρχομαι σε κάτι που είπαν οι προλαλήσασες. Στο θέμα της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας, αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία των Παρισίων και εξετάζοντας ε, ε, ενδελεχέστερα τις εθνικές υποσχέσεις συνεισφοράς που στηρίζουμε, αυτά τα, αυτές οι υποσχέσεις συνεισφοράς, οι ένδυσεις που προτείνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ πιο ευαίσθητες και συνεκτιμούν πολύ περισσότερο την ισότητα των φύλων από ότι οι αντίστοιχες ε, ε, ε, υποσχέσεις συνεισφοράς των βιομηχανικών, εκβιομηχανισμένων χωρών. Είναι πολύ εθαρρυντικό αυτό ότι συμπεριλαμβάνουν και την ισότητα των φύλων στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες και μάλιστα ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι άλλο που βλέπουμε στην αναπτυξιακή συνεργασία είναι ότι το θέμα των φύλων λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται και σε δραστηριότητες που αφορούν την προσαρμογή. Και αυτό που επιδιώκουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να μεριμνήσουμε ώστε η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου να λαμβάνεται υπόψη και στις δραστηριότητες για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Και μάλιστα στην ε, ΔΕΦΚΟ, στο ίδιο τμήμα που ασχολείται με τα τεχνολογικά θέματα και, και τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε ένα ειδικό τμήμα για την ενέργεια και, το, και την ισότητα των φύλων, ώστε ο τελικός χρήστης της ενέργειας ε, να συμβάλλει στη χειραφέτηση ε, του ανθρώπου και έτσι να μειωθούν οι ανισότητες και να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στην ανάπτυξη, να εξασφαλίζει το εισόδημά του και επίσης ε, να, ε, να σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα των αξιών και από τεχνική άποψη αλλά και από ηγετική άποψη ώστε να είναι όλοι αυτοί φορείς ε, αλλαγής. Κάτι που είναι σημαντικός παράγοντας για την πρόοδο. Αυτά και θα δώσω το, αφήσω το χρόνο για τις υπόλοιπες καλεσμένες. Η κυρία Δελτσότο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με ό,τι υπόθηκε για την συνέπεια συνεκτικότητα των πολιτικών. Φυσικά και είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα όσα πρέπει να έχουμε κατά νου. Σε ό,τι αφορά τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα, δεν είναι ένα ε, θέμα που αφορά των ελεγχογενήσεων αλλά αφορά την ευρύτερη πρόσβαση στην υγεία και υπό ορισμένες προϋποθέσεις ε, συνδέεται και με πραγματικές καταστροφές ε, όταν ε, εκτοπιστέντα άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πολλές φορές για τις γυναίκες εδώ τίθεται μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει και με τη βία και με πολλά άλλα ευρύτερα ζητήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you for being so... Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήσασταν και τόσο σύντομοι. Γιάννη Στέφανσον τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα και τα ζητήματα, τα πολύ σημαντικά που αναφέρατε. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω περαιτέρω είναι η ευθύνη που έχετε σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που παρέχετε. Έχει μεγάλη ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό. Και σε ό,τι αφορά το, το πράσινο κλιματικό ταμείο υπάρχουν πολλά χρήματα του ταμείου αυτού που ουσιαστικά ε, χρηματοδοτούν δράσεις που καταπατούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που γίνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ και που και αυτά καταπατούν τα δικαιώματα των αυτοκινήτων. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί και στη Σουηδία δεν έχουμε βρει ακόμη τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Και οι ΣΑΜΗ. εμεί ε, μπορούμε ε, να πούμε ότι εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας στο δικαστήριο. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, ούτε την νομική δυνατότητα όμως να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε μεγάλους ομίλους που παίρνουν αυτή τη χρηματοδότηση από το Green Climate Fund, για παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική και τις ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να διατηρηθούν. Μόνο στο προήμιο έχει περιληφθεί κάποια σχετική διάταξη, όχι στη συμφωνία ε, αυτή καθεαυτή. Αλλά πρέπει να βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες. Φαντάζομαι όμως ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να τα εξασφαλίσει αυτά. Ευχαριστώ η σε Ευχαριστώ πολύ και τώρα η Μέρι Ρόμπινσον για να κλείσει. Δεν είναι και τόσο Ηράκλειο το έργο σας. Από όλα αυτά που άκουσα, ε, τα πολύ ενδιαφέροντα από τις παρατηρήσεις, το θέμα της ε, ε, συνεκτικότητας και της συνοχής μας είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνέχεια σκέψης, ε, όχι όσον αφορά την σημασία της αλλαγής του συστήματος όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε και εύγλωτα αναφέρθηκε προηγουμένως χρειαζόμαστε κυκλική οικονομία βεβαίως αλλά πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Και αυτό που είπε η Χάιντι σχετικά με την ε, ε, καθαρή ανάπτυξη και το μηχανισμό Clean Development Mechanism. Ναι, έγιναν πολλά λάθη και νομίζω ότι τώρα ακριβώς γίνεται μια προσπάθεια διόρθωσης των λαθών αντιστροφής πορείας. Οπωσδήποτε πρέπει με μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε, ε, να επιβλέπουμε όλα τα μέτρα και όλους τους μηχανισμούς. Θα πρέπει να δούμε αυτούς ε, που παρέχουν καθαρή ενέργεια, εάν το κάνουν σωστά και αν σέβονται την ε, ισότητα των φίλων. Ξέρω από φίλους ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά παράπονα ε, και καταγγελίες ε, ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των γυναικών και την παραβίαση των αρχών αυτών από αυτούς που παρέχουν καθαρή ενέργεια πρέπει να ε, δουλέψουμε για το 1,5, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, ε, πρέπει, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, του θα είναι δύσκολα. Ε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε και όσον αφορά το μετριασμό και όσον αφορά την μετάβαση. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κατανοήσει πρώτα απ' όλα, ειδικά από εδώ και στο εξής, την ε, σημασία της διασφάλισης ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και της ισότητας των γυναικών. Όσον αφορά τις παρουσιάσεις που ακούσαμε από τις εισηγήτριες στο πάνελ, είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά που ακούμε. Βεβαίως αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ε, πρέπει να ενισχυθεί και η συνεργασία αλλά και η, και η χρηματοδότηση ε, θα πρέπει μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης να προωθηθεί ακριβώς έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η, αυτή η συμμετοχή στη βάση. Και όσον αφορά την ε, ε, όσον αφορά την θέση του νέου Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτιέρε ε, για το συγκεκριμένο θέμα και στα πλαίσια τη συγκεκριμένη επιτροπή για το Ελληνίνιο και οι προτάσει ε, που του κάνουμε είναι ότι θα πρέπει λίγο να βγούμε από τα εσκαμένα ε, Θα πρέπει ο καθένα να σπάσει λίγο του τείχου που περικλείουν τη σκέψη του και να βγει προς τα έξω ε, βεβαίως οι χώρες μας ε, θα πρέπει να παίξουν ηγετικό ε, ρόλο, θα πρέπει να είναι σε αυτήν την προσπάθεια. Πιστεύω ότι η έκθεση ε, την οποία ε, θα ε, ψηφίσετε για την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή και την κλιματική δικαιοσύνη πραγματικά θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής από μεμονωμένες χώρες. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι υπάρχει αναλογία με τον Τιτανικό. Όταν ο Τιτανικό σεισμός ε, χτύπησε στο παγόβουνο ε, δεν ε, πνίγηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους μονάχα αυτοί που ταξίδευαν στην τρίτη θέση, αλλά και αυτοί που ταξίδευαν στην πρώτη θέση και αυτοί που ήταν στο πιδάλιο. Επομένως, μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες, γιατί όλο και περισσότεροι θα είναι οι εκτοπισμένοι, όλο και περισσότεροι θα είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. ε, ακούω με μεγάλη προσοχή ε, το ψυχικό και ε, πραγματικό τραύμα της ε, κοινότητας των Σάμι. Ε, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τέτοιου είδους καταστάσεις γιατί εμείς θέλουμε μια νέα κλιματική οικονομία ε, η οποία θα στηρίξει τους πιο αδύναμους. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να δώσουμε προτεραιότητα στους τελευταίους που θα πρέπει να γίνουν πρώτοι θα πρέπει ακριβώς κατά προτεραιότητα να ασχοληθούμε ε, με τους πιο αδύναμους, με τους πιο τροτούς, με αυτούς που χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτή η έσχατη θα είναι η πρώτη και ότι ιδιαίτερα στις, αναπτυγμένες, στις αναπτυσσόμενες χώρες να βοηθήσουμε. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για οικογενειακό προγραμματισμό, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για στήριξη των γυναικών. Δυστυχώς έχει προκύψει τώρα και αυτό το νέο πρόβλημα του, του, του, αυτή η απόφαση για μείωση της χρηματοδότησης ε, των ε, ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων, αυτή η γενικευμένη απαγόρευση που μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει όμως, ε, στα δικά μας επιστρέφοντας, ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη χαρά ε, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και από την πλευρά του πάνελ και από τους αγορητές. Πραγματικά εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, κλιματική ποινική δικαιοσύνη και να δοθεί στις γυναίκες αυτός ο ηγετικός ρόλος που τους ταιριάζει και τους αρμόζει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρου ε, τη Επιτροπή των Γυναικών, τη Μέρι Ρόμπινσον και όλε τι καλεσμένε του πάνελ ε, για την έμπνευση που μα έδωσαν με τι προτάσει του. Και τώρα η συγκεκριτρία. Ναι, πραγματικά είμαι συγκλονισμένη. Ε, πραγματικά με εμπνεύσατε και με ψυχώσατε. Θα ήθελα να πω κάτι για την ηθαγένεια και την ενεργό ηθαγένεια, γιατί είναι και αυτό συναφές θέμα. Και ευχαριστώ, Τζάνι, που μίλησες τόσο σταράτα, ε, τόσο συγκινησιακά φορτισμένα. Ήσουν πραγματικά καταπληκτική και πραγματικά θερμά συγχαρητήρια. Άγγιξες ε, την καρδιά μου πραγματικά με αυτά που είπες. Ε, και όπως είπε η Μαρία Ράπης, θα πρέπει να γίνουμε δέσμοι της ελπίδας, ε, να ακούσουμε τις άλλες φορές να να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και να υψώσουμε στα δόρια τη φωνή των γυναικών. Έχουμε τώρα μια αντιπροσωπή από τη Σουηδία που δεν ε, συμμετέχει σε πολιτικό κόμμα και είναι πραγματικά δέσμοι τη ελπίδα. Μπορείτε να σηκωθείτε γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή σα. Θα μπορούσα να είχα συντάξει και μόνη μου την έκθεση, αλλά πραγματικά ε, χρειαζόμαστε δραστήριου πολίτε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με την ελπίδα του στον νόμο και ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτή τη δημόσια ακρόαση. Είστε πραγματικά πολύ σημαντικοί για μένα. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα και βλέπω στην ομίγυρη αρκετούς ευρωβουλευτές αλλά περισσότερους καλεσμένους εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα βάλουμε την έκθεση αυτή και στο σύστημα, αλλά θα την προσπαθήσουμε να τη διαδώσουμε. Θα τη διαβάζει η Μέρη, ε, η Μέρη Χάνιμπολ, αλλά εσείς ε, θα πρέπει να μας, βοηθήσετε, εσείς να βγείτε στο δρόμο με τις οργανώσεις σας σε όλα τα επίπεδα ε, της κοινωνίας και να ε, μιλήσετε για τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της συνεδρίασης. Ευχαριστώ και πάλι τους καλεσμένους. Παρακαλώ πρέπει να συνεχίσουμε γιατί η ώρα περνάει. Και σε τέσσερα λεπτά κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, κάτι που μάλλον απίθανο το βλέπω. Ας ε, εξετάσουμε όμως το σημείο 6 πρώτα, τα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ε, δράσεις για τον προϋπολογισμό του 2018 η συγγήτρια είναι η Κωνσταντς Λεγκρίπ, η οποία όμως απουσιάζει, οπότε θα την αντικαταστήσει η κυρία Γκάρ Πέλτς. Παρακαλώ, κυρία Γκάρ Πέλτς, κάντε μας ε, μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης Λεγκρίπ, γιατί όπως σας είπα έχουμε μείνει πολύ πίσω στο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την κυρία Λεγκρυπ που κολλείεται σήμερα θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε τα προγραμματικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές ε, δράσει για το 2018. Θα υποβληθεί στην Επιτροπή Προπολογισμού και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την, ε, την διαδικασία για τον προπολογισμό. Εννέα είναι τα δοκιμαστικά σχέδια από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή μας. Έτσι έχουμε ένα ευρύ φάσμα προτάσεων που καλύπτουν θέματα ενδιαφέροντος όπως γυναίκες και χρηματοδοτικό πλαίσιο, χειραφέτηση των γυναικών εργαζομένων. Η κυρία Λεγκρύπ εξέτασε τα σχέδια που υπευλήσα στη γραμματεία και προτείνει μια αξιολόγηση αυτών. Κατέληξε μάλιστα σε κάποια συμπεράσματα για τα προτινόμενα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις, τα οποία θα θα σα παρουσιάσω εδώ. Η κυρία Λεγκρίπ επισημαίνει το γεγονό ότι μερικά σχέδια 1, 2 και 3 είναι συνεπή, εφικτά και προτείνουν αποτελεσματικές δράσεις και μάλιστα ε, ξέρει το πολύ σοβαρό και αξιόλογο έργο που κατέληξε στην τα τρία αυτά δοκιμαστικά σχέδια και θα την Επιτροπή να τα υπερψηφίσει. Επίσης, θεωρεί ότι οι μελέτες που παρουσιάζονται στα σχέδια 4 και 8, παρόλο που προϋποθέτουν σημαντικές δαπάνες, ίσως ε, αποφανούν πολύ χρήσιμα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσχολικής εκπαίδευσης ε, παιδιών σε, στην ανεργία γυναικών από πολλούς τομείς. Επίσης, η κυρία Λεγκρίπ τη, τα μέλη της Επιτροπής να υπερψηφίσουν αυτά τα δύο σχέδια, 4 και 8. Παρ' όλα αυτά, με λύπη της, ε, η κυρία Λεγκρίπ κρίνει ότι τα προγράμματα 5, 6 και 7, παρόλο που δυνητικά θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, δεν είναι αρκετά ακριβή και σαφή, οπότε σας ε, προτείνει να τα καταψηφίσετε. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο 9, η κυρία Λεγκρίπ ε, θεωρεί ότι το σχέδιο 9 που θέλει να εφαρμόσει συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεν αποτελεί κατάλληλο εργαλείο. Θεωρεί ότι εναπόκειται στα, κρα... στα κοινοτικά θεσμικά όργανα να προσδιορίσουν τις πολιτικές συνεκτίμησης της διάστασης ε, φύλου. Οπότε δεν είναι λόγος ε, να τις θέσει η Επιτροπή σε διοργανική βάση και στο πλαίσιο μάλιστα μιας ε, προπαρασκευαστικής δράσης. Γι' αυτό το λόγο η κυρία Λαγκρή φτάσεται κατά του σχεδίου 9. Μετά την ψηφοφορία για τα πιλωτικά αυτά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις θα κατατεθούν πριν τις 3 Μαΐου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για προαξιολόγηση, προκατακτική αξιολόγηση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα λάβουμε και την ε, ε, προαξιολόγηση στα τέλη Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την ανταλλαγή απόψεων που θα γίνει τον Ιούλιο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα προχωρήσει το θέμα. Η κυρία Λεγκρίπαση ε, ευχαριστεί θερμά ο συνέβαλα στην υποβολή των προγραμμάτων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων και σας προτείνει να ακολουθήσετε τις συστάσεις και επίσης προτείνει να δοθεί ευκαιρία στους συναδέλφους να υποβάλουν πιο λεπτομεριακές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαλπέλτς, εκ μέρους κυρίας Λεγκρυπ. Θα έχουμε τώρα σύντομες παρουσιάσεις από όσου κατέθεσαν αυτά τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. PP1, στοχευμένες δράσεις για την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Σύρπα κάνανε η εισηγήτρια. Η συγγήτρια Λαγκρή προτείνει να υπερψηφίσουμε αυτό το θέμα, αυτό το σχέδιο. Δεύτερο ε, πιλωτικό σχέδιο, η βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία της μητρότητας για τις ευάλωτες ομάδες. Μαρία Ρενά. Νομίζω ότι είναι εύγλωτος ο τίτλος. Θέλουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγεία των μητέρων γιατί διαπιστώνουμε μία διάκριση βάρος των ευάλωτων ομάδων. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν που βρίσκονται στενοποίοι του προβλήματος ε, και αν μπορούμε να έχουμε μετά ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ένα, περισσότερα μέτρα ορθολογισμού, κυρίως προς τις ευάλωτες ομάδες που θίγονται περισσότερο από αυτό το πρόβλημα, την ελληνική πρόσβαση στην υγεία. Ε, δοκιμαστικό ε, σχέδιο 3 ε, η χειραφέτηση των κοριτσιών στον κόσμο. Μπεατρή Μπεσέρα, Εσταρά Φεραγκούτ. Ποιος, ε, ποια είναι παρούσα. Ευχαριστώ, λέει, κυρία Μπεσέρα. Θέλω να σα ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε, που μα δίνετε τη δυνατότητα να σα μιλήσουμε για την πρόταση αυτή για να δώσουμε τη δύναμη στις αυριανές ηγέτιδες ε, Δυστυχώς ε, εξακολουθούν να υπάρχουν ε, οι ανισότητες ε, στην κοινωνία μας. Περιορίζονται οι φιλοδοξίες των νερών κοριτσιών και από πολύ νεαρή ηλικία μειώνονται οι επιλογές τους. Άρα η καλύτερη ιδέα εμείς να κάνουμε τη διαφορά και να αλλάξουμε αυτές τις πραγματικότητες είναι να πετύχουμε κάποιους βασικούς στόχους, δηλαδή για, τις, για τα κορίτσια από 10 έως 15, να έρθουν αντιμέτωπες με διάφορες θέσεις εργασίας, να δουν διάφορα μοντέλα μοντέλα, διάφορες ρόλους και υποδείγματα, να δώσουμε έμπνευση στα κορίτσια. Δεν θέλουμε να τους επιβάλλουμε κάποια μοντέλα, απλά να τους ε, τα παρουσιάσουμε, ε, να δουν τα διάφορα υποδείγματα, τα διάφορα καλά παραδείγματα που υπάρχουν ε, από εκτελεστικά στελέχη, ε, τις ε, γυναίκες που απασχολούνται σε μερική μόνιμη απασχόληση κτλ. Θέλουμε επίσης να σπάσουμε τα στερεότυπα και τους παραδοσιακούς ρόλους και μοντέλα. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα νομίζω ότι συμπληρώνεται και το θέμα της χρηματοδότησης και της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σημειώστε το παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, αυτή είναι σωστή διατύπωση και υπάρχει θετική νομίζω αξιολόγηση για αυτό το πρόγραμμα. Περνάμε στο 4 τώρα. Πώς επηρεάζει η φτώχεια, για παράδειγμα, της οικογένεια και τα Κύριος Πιμέντα Λόπες ε, καταθέσει αυτό το project. Δεν είναι εδώ. Θα ήθελε κάποιος άλλος να παρουσιάσει το θέμα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μήπως λοιπόν θα ήθελε κάποιος συνάλφος που είναι ε, τον, για όλα για τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα να μας τα παρουσιάσει συνοπτικά. Όχι. Άρα πάμε στο 9, το τελευταίο. Για την ε, σωμάτωση της διάταξης του φίλου στη, στα θεσμικά όργανα, ο Ερνέστ Ουρτασούν. Ε, ναι, ευχαριστώ. Να στηρίξετε παρακαλώ αυτό το project για να υπάρχει ένα συντονισμό τη διάσταση ε, του φίλου, συμπερίληψη διάσταση του φίλου σε όλα τα θεσμικά όργανα τη Ένωση. Νομίζω ότι ο προβολισμό είναι περιορισμένο. Θα ήταν καλό λοιπόν να δούμε πώ γίνεται αυτό το gender mainstreaming. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που σας έβιασα λίγο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, ελπίζω να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το ορίζοντα 2020 καταρχάς και τα πιλωτικά προγράμματα. και την ακαδημαϊκή ε, και εξαποστάσεω εκπαίδευση στο πλαίσιο τη αντίκηση για τη διαβίου μάθηση. Λοιπόν, αξιολόγηση το ορίζοντα 2020 είναι το πρώτο θέμα που θα ψηφίσουμε. Αξιολόγηση τη υλοποίηση του προγράμματο με γνώμη την διάμεση αξιολόγησή του και την πρόταση για το το πρόγραμμα πλαίσιο. Η συγκέντρα δεν είναι εδώ, άρα δεν μπορεί να πει τίποτα. Επομένω, πάμε στη συμβαστική 6. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 24 καταπίπτει. Πηγαίνουμε στην 16. Ψήφι υπέρ κατά, κατά απορρίπτεται 17 υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται, τροπολογία 5 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε παρακαλώ αμφίροπον το αποτέλεσμα. Voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Μία ψήφος διαφορά εγκρίθηκε. Συμβαστική 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το ελέγξω όμως. Ηλεκτρονικά για την 8, τη συμβιβαστική. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. 29. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, όχι. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, Ορίστε, τι είπατε. Συγγνώμη, δεν έχω την πιο επικαιροποιημένη λίστα ψηφοφορίας. Τέλος πάντων, καλά τα έλεγα εγώ, τροπολογία 51, ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 10, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα πάμε στη συμβαστική 11, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα είμαστε στην τροπολογία 41 και τη 44 που είναι ταυτόσιμε ψήφι υπέρ. Κατά. Αγκρίνονται. 42 ψήφι υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ψήφι περ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 50. ψηφι περ. υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 52-53 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στις ετυλικές σκέψεις. 1. Υπέρ, κατά, ποιες, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, τροπολογία 6, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Νομίζω ότι τώρα Ήρθε η ώρα για την τελική ψηφοφορία, η οποία θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Επόμενο θέμα και επόμενη ψηφοφορία. είναι τα πιλωτικά προγράμματα. Ε, παράγραφος, ε ε, ε, ε, ε, συγγνώμη, πιλωτικό πρόγραμμα 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 2 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 3. Υπέρ. Α, ε, επί του 3 υπάρχει μια προφορική τροπολογία της κυρίας Μεσέρα. Θέλετε να παρουσιάσετε μήπως την προφορική σας τροπολογία. Στην ουσία αφορά μία διόρθωση του τίτλου Empowering Girls in Europe αυτή είναι η διόρθωση. Θέλουμε in Europe, στην Ευρώπη και όχι στον κόσμο, around the world. Ωραία, εξαιρετικά. Πιλωτικό πρόγραμμα 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 5 λέει η πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αυτό απορρίπτεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται επίσης. Πιλωτικό πρόγραμμα 7. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 8. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Πιλωτικό πρόγραμμα 9 υπέρ κατά. Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Περνάει και αυτό. Με διαφορά μιας ψήφου, αλλά πάντως περνάει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και για αυτή την ψηφοφορία. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Τελευταία λέω. Αφορά την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και ως εκπαίδευση ως μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διαβίου Μάθηση. Τροπολογία 13, γιατί έχει αποσυρθεί 14, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15. Α, όχι, καταπληκτή 15. 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Όχι, 19. 19 διορθώνει πρόεδρος υπέρ. Κατά. Περνάμε τώρα στην 20. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Δεν είμαι σίγουρη. η Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. κατά τμήματα, κατά δύο τμήματα. Έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ε, κατά τμήματα δηλαδή, υπέρ, κατά, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά α, εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά Νομίζω πως απορρίπτεται. Ναι, απερίφθη. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 32 όχι, 33. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά εγκρίνεται επίσης. Και αυτή ήταν η τελευταία μας ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Okay, Σας ε, ευχαριστώ όλους όσοι παρέμειναν για το τέλος της συνεδρίασης. Θα χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου για να βάλω λίγη τάξη. Τάξη, όπως λένε και στη Βουλή των Κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημείο 6 οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Άννα Χέντιν, η συγκεκριά μας, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ταξομίκε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσής μου. Προς το παρόν έχει τη μορφή εγγράφου εργασία. Όπως ξέρετε, θέμα της έκθεσης είναι η οικονομική χειραφέτηση ή ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ευρύτατος ε, τίτλος, ε, αρκετά γενικός και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε το θέμα από διαφορετικές κοπιές και πρίσματα. Γι' αυτό και στο έγγραφο θα έχω αρκετές προτάσεις. Ε, έγινε ήδη μια πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και μετά την ανταλλαγή απόψεων ελπίζω το σχέδιο έκθεσης να σας ε, ε, αφήσει ικανοποιημένου, αλλά όσοι έχουν να υποβάλουν προτάσεις περαιτέρω και τροπολογίες ε, είναι ευπρόσδεκτοι. Μερικές προτάσεις είτε είναι υπερβολικές, είτε αφορούν εθνικές αρμοδιότητες και όχι κοινοτικές, οπότε είναι εκτός θέματος. Πάντως, όλοι είμαστε στρατευμένοι υπέρ της ενίσχυσης της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέρ της ε, ε, ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών. Οπότε, να πω και σε εμά ε, ως ερετούς και ως εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών να απευθύνουμε εκκλήσεις στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μέτρα και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση μιας πραγματικής ισότητας. Αυτό είναι το καθήκον μας. Και εξού και ε, οι απαιτήσει μου στην έκθεση να έχουμε μια χαρτογράφηση της διαμόρφωσης των, των μισθών και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι θα έχουμε καλύτερη επίγνωση κατάσταση και θα εντοπίσουμε τους ε, μη αντικειμενικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τους μισθούς, ε, ώστε να καταλήξουμε σε ισότιμα ή σε επίπεδα μισθών. Ε, αυτό ενδιαφέρει λοιπόν τους εργαζομένους και κυρίως τις γυναίκες. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε την κατάλληλη προσέγγιση και τα εργαλεία, ώστε να αναβαθμίσουμε κάποιες θέσεις γιατί μέχρι στιγμή οι ενδοκρατούμενε ε, θέσει εργασίας θεωρούνται πιο αξιόλογες. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, να αναδείξουμε την αξία και άλλων κατηγοριών ε, εργασιών που είναι ίσως πιο γυναικοκρατούμενες προς το παρόν και να συμβάλλουμε σε μια πιο ακριβοδίκαιη διαμόρφωση των μισθών. Θα λάβω υπόψη τα σχόλιά σας, ώστε να διευρύνω την έκθεση. Μερικοί μίλησαν για κατάρτιση και εκπαίδευση των γυναικών και στηλίτευσαν το θέμα της ε, βίας εις βάρος των γυναικών. Ένα είδος βίας είναι και η οικονομική βία, η οικονομική εξάρτηση των γυναικών που απειλεί την ε, ελευθερία τους, ακόμη και την ίδια την επιβίωσή τους. Επίσης, ε, η έκθεση αφορά την ε, οικονομική κατάσταση των γυναικών και την οικονομική αδικία δυστυχώς που διέπει πολλές φορές τη ζωή τους. Πάντως προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τους κοιόδης ηγητέ και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές γιατί δυνάμεθα και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να καταστήσουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ε, χώρο που θα απολαμβάνουν ισότητα οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης, ε, εισηγήτρια, γι' αυτό θα ήθελα εκ μέρους του να αναφέρω τις σκέψεις μας. Η ε, κυρία Γκαλπέλης, καταρχάς συγχαίρω την κυρία Χέντ για την έκθεσή της. Ήταν ε, πολύ αποτελεσματική εργασία της και νομίζω ότι το σχέδιο έκθεσης είναι καλό. Και εγώ προσωπικά συμφωνώ με το περιεχόμενό του, γιατί πιστεύω ότι η έκθεση συμμορφούνται πλήρως προς την αρχή της επικουρικότητας. Ο ρόλος των γυναικών και η οικονομική τους χειραφέτηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι γυναίκες είναι μια σημαντική πηγή, ένα σημαντικός πόρος της κοινωνίας. Αν δεν του δώσουμε του πόρου αυτού τη δέουσα προσοχή, θα είναι σε βάρος μας. Είναι θέμα ανταγωνιστικότητας ουσιαστικά και ισότητας βέβαια. Η αύξηση της γενικής απασχόλησης ε, και η μείωση της ε, ανεργίας ή αδράνειας ε, είναι κάτι που θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις. Κοινωνικές υπηρεσίες όπως είναι η παιδική μέρημνα, η φροντίδα των ηλικιωμένων απαιτεί νέα μοντέλα, νέα σκέψη οι γυναίκε δεν θέλουν να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της οικογένειάς του ή της εργασίας. Ε, θεωρούν και τα δύο είναι σημαντικά. Η σταδιοδρομία τους είναι εξίσου σημαντική με την οικογένειά τους. Έτσι πιστεύουν. Σε ό,τι αφορά την αρχή της ίση αμοιβή για ίση εργασία, για την ίδια εργασία, το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν μπορούμε να θέτουμε αυθαίρετες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αρχή της ίσα ε, για την διαργασία ήταν καθαρά οικονομικό το θέμα και στη νομοθεσία προς το παρόν προβλέπονται μόνο μη δεσμευτικά μέτρα για τις χώρες μέλη. για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι αμοιβέ, οι ε, μισθοί δεν είναι ευσεβείς πόθη, είναι, έχει να κάνει με την λειτουργία της οικονομίας και, της οικονομικής, και την οικονομική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πολιτικές στην Ευρώπη που θα οδηγήσουν σε ισοτιμία μισθολογική και μεταξύ των και γυναικών αλλά και μεταξύ κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι άλλο σημαντικό. Ναι, μεν σήμερα οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση και έχουν μάλιστα και καλύτερες επιδόσεις ε, στατιστικά. Τι βλέπουμε, ότι οι γυναίκες παίρνουν 25% λιγότερο και υποεκπροσωπούνται στις διοικητικές θέσεις. Άρα πολλά απομένουν να γίνουν. Άρα μπορούμε να διατυπώσουμε συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Θα καταθέσω τροπολογίες που ελπίζω να προσφέρουν στη θέμενη αξία. Ουσιαστικά μιλάμε για μια οικονομική προσέγγιση. Έχουμε όμως και τα θέματα της βίας σε βάρος των γυναικών. Και δεν θα πρέπει να δούμε τα καθημερινά φαινόμενα βία. Ε, ε, έχουμε τη βία στον τόπο εργασία. Επίση αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε στις γυναίκες περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εκπαίδευση και στην ψηφιακή εκπαίδευση και στη διαβιομάθηση. Μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Είναι καλή έκθεση, είναι καλή αφετηρία για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Οι επόμενη, επόμενες ε, να είναι σύντομοι διότι είναι ήδη εξ και τέταρτο. Από την ομάδα ECR, κύριε Βυσνιέσκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ως ε, ε, και όλες τις στα θέματα αυτά οικονομικής χειραφέτηση των γυναικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγητρία για την εκπόνηση του σχεδίου έκθεση και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων για ένα έγγραφο που περιλαμβάνει βασικές απόψεις προς τις οποίες συμφωνούμε. Νομίζω ότι ε, είναι αυτονόητο ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών όχι μόνο είναι κάτι που όχι μόνο είναι δίκαιο αλλά και έξυπνο, ευφυές. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την ιδέα. Η οικονομική ενίσχυση των γυναικών θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και αποτελεσματική. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε δίκες, έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Ε, γιατί οι γυναίκες αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα που επισημαίνονται πολύ εύστοχα στην έκθεση και χαίρομαι που η συγγήτρια ε, κατά προτεραιότητα αναφέρει τα προβλήματα των ε, γονιών που προσπαθούν να εξορροπήσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική του ζωή και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε νέες δυνατότητες ε, εργασίας και απασχόλησης και να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα είναι η ε, ίση αμοιβή για ισότιμη εργασία και για τις γυναίκες ε, και επίσης ε, ίσες συντάξεις. Η Πολωνία πρωτοστατεί στα θέματα αυτά και μάλιστα έχουμε θετικά αποτελέσματα χωρίς ρηξικέλεθες μεθόδους. Επίσης για να έχουμε κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να κάνουμε σωστή διάγνωση της, του ιατρικού προβλήματος. Ε, δεν συμφωνώ απόλυτα εδώ με την εισηγήτρια, γιατί το να ε, αποδίδουμε όλα τα προβλήματα των γυναικών σε παραδοσιακά στερεότυπα είναι μια εύκολη λύση, αλλά δεν είναι πάντα ε, σωστή και μερικές φορές μας οδηγεί και σε σφαλμένα συμπεράσματα. Γιατί η ισότητα και η ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης είναι απαραίτητη, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε μείωση των ικανοτήτων τους, γιατί πραγματικά οι γυναίκες ούτε ε, είναι λιγότερο έξυπνες, ούτε λιγότερο ικανές από τους άντρες. Θα ήταν λάθος να σκεφτεί κα, κανείς ότι με, με τεχνική ισότητα θα έχουμε μια δημοκρατική νομοποίηση των δημοσίων φορέων. Νομίζω ότι εκφεύγουμε εδώ από το περιεχόμενο της συνθήκης. Επίσης, ε, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και τις γυναίκες που μόνος ανατρέφουν τα παιδιά τους και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παιδιών. Για όλα αυτά τα θέματα θα καταθέσω τροπολογίες και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε με αγαστή συνεργασία να διαμορφώσουμε μια πολύ αξιόλογη έκθεση και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πιστεύω θα είναι καρποφόρα η συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Η Μόνικα Βάνα έχει το λόγο από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά την συγκίτρια την κυρία Χέντ για το σχέδιο έκθεση που υπέβαλε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι που αποτελεί καλή βάση για συζήτηση και συμφωνώ με τα περισσότερα σημεία της έκθεσης. Βέβαια, δεν θεωρούμε ότι εξαντλείται όλο το φάσμα των ε, θεμάτων που είναι συναφή με, με την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Βέβαια, τα ουσιώδητα καλύπτεται και συμφωνούμε ότι η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς Συγγνώμη, έχει κλείσει το μικρόφωνο της ε, κυρίας Βάνα. Τι έγινε, συγγνώμη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το θέμα της οικονομικής χειραφέτησης έχει κέρια σημασία και για τη μείωση των ανισοτήτων και για την υλοποίηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Και οι τομείς όπου θα καταθέσουμε τροπολογίες είναι η εξή. Καταρχήν θα πρέπει να, να αναφερθούμε στο πακέτο εξορρόπηση ε, του προσωπικού και επαγγελματικού βίου. Αύριο θα υποβάλει το τη σχετική Δεσμημέτρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω το δικαίωμα στην άδεια πατρότητα και τη ε, μη φορητότητα τη της ε, γονική άδεια. Νομίζω στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να αποκρισταλώσουμε τη γνώμη μας. Ό,τι αφορά την παράγραφο για, την, για τον ίσο μισθό, να αναφέρουμε το θέμα των, ελάχιστων, των κατώτατων μισθών και την αξιοπρεπή απασχόληση. Νομίζω αυτή είναι βασική στόχη για την υλοποίηση ισότητας και ίσης αμοιβή. Επίσης, το θέμα της βίας. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόνο στο αρχικό επεξηγηματικό σημείωμα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το οικονομικό κόστος της βίας, να έχουμε ένα σχετικό εδάφιο. Επίσης, μιλούμε για, κυρίως για το δημόσιο τομέα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και σημαντικό για τις γυναίκες. Ε, η εξασφάλιση δημοσίων υπηρεσιών για τις γυναίκες επίσης θα πρέπει να αναφερθεί. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 61η συνέλευση ε, των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ε, στην οποία είχαμε λάβει μέρος, ε, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί στην έκθεση. Θα καταθέσουμε τροπολογίες για δείκτες για τη συνεκτίμηση των φύλων, για την εκπαίδευση, ποσοστώσεις, ενεργειακή ένδυα, εργαζόμενες στην Ήπεθρο και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστριών και γυναικών προσφύγων. Αυτά προς το παρόν, να και ο χρόνος είναι περιορισμένος και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ε, λέει η κυρία Γιούτο, γιατί ε, πραγματικά έχει επιλέξει μια ικανοποιητική ε, κίνηση ε, που μας βρίσκει σύμφωνος ε, σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως αυτή η προβληματική θα πρέπει να λυθεί, που δεν θα ολοκληρωθεί βεβαίως η αντιμετώπιση ε, του προβλήματος και θα λύσει το πρόβλημα ε, αυτή η έκθεση, ωστόσο θα αποτελέσει μία ακόμα πίεση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ενδεχομένως ε, θα αποτελέσει κίνητρο έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως κατανοούμε ότι δεν αρκεί να επιβληθεί μέσω νομοθεσίας ε, η ισότητα των μισθών γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες διαθέτουν νομοθεσία ισότητας των φύλων αλλά δεν εφαρμόζεται. Ε, το ίδιο ε, συμβαίνει όπως και σε άλλες περιπτώσεις και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Βεβαίως εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν καλοί νόμοι για την ε, ισότητα των αμοιβών. Αλλά εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε αυτοί οι νόμοι ε, να εφαρμοστούν πραγματικά, να βρουν αντίκτυπο στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητα των γυναικών ε, στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα όπως ας πούμε είναι η βία κατά των γυναικών σε πολλές χώρες. Υπάρχει νομοθετικό πλωστάσιο εξαιρετικό. Ωστόσο, επιτόπου που ε, ε, υπάρχει μεγάλη διάσταση ανάμεσα ε, σε αυτά τα ωραία που είτε γράφουμε εμείς είτε περιλαμβάνονται στους νόμους και του τι συμβαίνει επί τόπου. Εμείς θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες αλλά πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο η συγγήτρια αντιμετωπίζει το θέμα και σαφώς πιστεύω ότι ακολουθεί την κατεύθυνση την οποία και εμείς επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ αργά και έχουμε ακόμα ένα θέμα με εξωτερικό ομιλητή. Θα ήθελα να ε, παρακαλέσω την εισηγήτρια, εάν συμφωνεί, να μην απαντήσει η ε, διερμηνής. Ε, μας παραχώρησαν πέντε επιπλέον λεπτά. Πολύ σύντομα, αν θέλετε. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζετε ότι το θέμα είναι ευρύ και δεν έχουμε βεβαίως τον χώρο έτσι ώστε να βάλουμε όλα τα θέματα. Χαίρομαι, πολύ ε, για τις ωραίες ιδέες που ακούω ότι έχετε. Γι' αυτό λοιπόν σας παροτρύνω ε, να υποβάλλετε τροπολογίες γιατί εμείς θα έχουμε με τον τρόπο αυτή την ευκαιρία να εκφράσουμε πραγματικά τις απόψεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ε, εργασία που έχετε κάνει. 12 ε, Μαΐου είναι η προθεσμία, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο μας ε, θέμα. Είναι η επίσκεψη του Ιδρύματος Καβίνα Τιλ Καβίνα ε, του Ιδρύματος αυτού και προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε την ομιλήτρια που μόλις έφτασε. Είναι η κυρία Πεσεύσκα. Τη ζητήσαμε να έρθει γιατί η Επιτροπή μας θα οργανώσει τον Ιούνιο μία κοινή διοργάνωση Για τις ε, χώρες διάβρισης και η ε, κυρία Μπασένσκα ε, θα μιλήσει για τα Δυτικά Βαλκάνια, κυρίως δε για τον περιορισμό του χώρου, τη συρρήκνωση της κοινωνίας των πολιτών και τα προβλήματα των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Γυναικών. Εμείς εκπροσωπούμε ε, έξι χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων και θα, θέλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις τελευταίες εξελίξεις των δικαιωμάτων των γυναικών. Στη δεκαετία του 90 ε, ε, άλλαξαν οι καταστάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Διαβρύνθηκε ε, η έλλειψη ισότητας όσον αφορά τις ευκαιρίες ανδρών και γυναικών έγιναν προσπάθειες βελτίωσης της θέσης των γυναικών, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν τα προβλήματα να είναι μεγάλα οικονομικές, ε, η οικονομική πραγματικότητα στις χώρες αυτές δεν δίνει την ε, δυνατότητα στις γυναίκες να αναπτύξουν τις οικονομικές ε, δραστηριότητες. Η κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι γυναίκες θίγονται, πλήγονται περισσότερο από την φτώχεια. Οι γυναίκες κατά 40% ε, βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας γυναίκες ε, ε, σε ηλικία ενεργή. Πολύ ε, συχνά επίσης ε, στις γυναίκες που εργάζονται σε βιομηχανίες έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παραβιάσεων των ε, εργασιακών τους δικαιωμάτων. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες έχουν μείνει εκτός της αναπτυξιακής διαδικασίας, της οικονομικής διαδικασίας, πράγμα που αποτελεί τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Έχει αυξηθεί ε, η ε, εκπροσώπηση των γυναικών στις, ε, στα κοινοβούλια. Είναι περισσότερες δηλαδή οι γυναίκες βουλευτές στα κοινοβούλια. Ωστόσο, όσον αφορά τις υψηλόβαθμες θέσεις, διαδικασία λήψεων αποφάσεων, θέσεις υπουργών κτλ. Ακόμα είναι λίγες οι γυναίκες οι οποίες παίρνουν τις θέσεις αυτές. Ε, επίσης ε, οι γυναίκες δεν παίζουν ε, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επίλυση κρίσεων που έχουν αντιμετωπίσει οι χώρες αυτές ή αντιμετωπίζουν τώρα. Σύμφωνα και με το ψήφισμα 2025 των Ηνωμένων Εθνών, οι γυναίκες δεν έχουν παίξει ε, σημαντικό ρόλο στις ε, διαδικασίες και τις ε, διαπραγματεύσεις στην Σερβία ή στο Κωσυφοπέδιο. Στο Μαυροβούνιο και το, την Φύρομ δεν φαίνεται καθόλου να παίζουν ρόλο οι γυναίκες στις διαδικασίες. Ε, η ε, μη συμμετοχή των ε, γυναικών στις διαπραγματεύσεις αυτές και τις πολιτικές διαδικασίες περαιτέρω δυσκολεύουν την θέση των γυναικών στις χώρες αυτές. Ορισμένες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων περιορίζουν τα σεξουαλικά δικαιώματα και τα δικαιώματα αναπαραγωγής των γυναικών κυρίως όσον αφορά ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως είναι η Ρωμά. Ε, ορισμένες από, ε, ορισμένοι από τους πρόσφατους νόμους ε, κατά το, την έννοια αυτή είναι ακόμα και αντισυνταγματικοί. Ένα άλλο θέμα που μας προβληματίζει περισσότερο είναι το κράτος δικαίου κυρίως ε, λαμβάνοντας ε, υπόψη τα περιθώρια που αφήνει ο νόμος όσον αφορά την ε, βία βάση του φύλου. Σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχεται ούτε η ελάχιστη προστασία μεγάλου αριθμού πολιτών. Το νομοθετικό πλαίσιο για την οικογενειακή βία ακόμα ιστερεί. Ε, οι χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων καταγράφουν πολλές ε, περιπτώσεις δολοφονιών γυναικών έστω και εάν οι γυναίκες είχαν προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσουν την, τις αρχές πριν την δολοφονία τους. Είναι περιορισμένη επίσης αν ε, εφόσον υπάρχει έστω και σε μικρό βαθμό ε, η ε, κρατική χρηματοδότηση που θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες. Επίσης η πρόσβαση σε υπηρεσίες είναι περιορισμένη για τις γυναίκες. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα συνολικά στα Δυτικά Βαλκάνια θα αναφερθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα. Επιθέσεις και ε, ε, κατηγορίες από την ε, πλευρά των αρχών χωρίς η συγκεκριμένη αναλυτική διαδικασία, καταχρηστική οικονομική έλεγχη ε, έλεγχη στις ε, μεγάλες και κυριότερης ε, σημασίας οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δυσκολεύεται όλο και περισσότερο η διαδικασία διαβούλευσης. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά παρόλα αυτά δεν δίνεται λόγος στις σε οργανώσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες ε, διεύρυνσης. Εάν ε, δεν ληφθεί υπόψη και η διαδικασία και η, η, διάσταση του φύλου στις ε, ε διαδικασίες, τότε δεν θα μπορέσουν οι διαδικασίες αυτές να ολοκληρωθούν ε, επιτυχώς. Πιστεύουμε ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι σημαντικό για την ε, για τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, ε, πιστεύουμε ότι εσείς είσαστε οι φυσικοί μας σύμμαχοι και στρεφόμαστε προς εσάς για βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε τα Μαρία Μπασέφσκα που ήρθε εδώ και μας μίλησε. Μας έκανε αυτή την επισκόπηση της κατάστασης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Λυπηρό μεν, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε χρόνο για συζήτηση. Λυπούμε πολύ, αλλά ήταν πολύ φαρτωμένη η μέρη διάταξη τη Επιτροπή μα και οι ερμηνείς δεν μπορούν να δουλέψουν περισσότερο. Η Τζούλη, παρακαλώ. Um, I'm one of the MEPs who's on... Είμαι μία από τι ε, βουλευτέ που είμαι μέλο αντιπροσωπεία για τι σχέσει ε, με Βοσνία-Ζεγοβίνη Κοσμοπέδιο και ήμουν ε, την προηγούμενη εβδομάδα εκεί σε σχέση με την κοινή, μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση τη Συμφωνία Σύνδεση και έχω επαφές με τις ε, εθνικές οργανώσεις ε, εκτός κοινοβουλευτικής ε, δράσης μου. Συναντηθήκα με πολλές γυναίκες σε διάφορα κέντρα και πήγα και σε μια από τις πόλεις που δεν ξέρω αν την προφεκάω, τέλο πάντων είχε πάρα πολλά θύματα σεξουαλικής βίας στη δέκα του πολέμου. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να συζητήσει την κατάσταση των γυναικών σε αυτές τις χώρες που έχουν βιώσει τέτοια καταστάσεις χωρίς να μιλήσουμε ακριβώς για αυτά τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την ε, ευημερία τους, με την ονομική τους ευημερία. Με τις γυναίκες που μίλησα ε, μου έλεγαν ότι δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν καμία αποζημίωση και επειδή δεν, έχει απο... δεν τους έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, εξακολουθούν να φέρουν τραύματα 18 χρόνια μετά τον πόλεμο. Νιώθουν ότι δεν έχει αποκατασταθεί αδικία δεν έχουν ξεπεράσει τα τραυματά του. Και είναι πολύ σημαντικό μέρη που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά νομίζω θα πρέπει να δείξουμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει κάποιε από τι βασικέ αιτίε που αποτρέπουν τι γυναίκε από το να ε, αναπτύξουν εντελώ το δυναμικό του στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων ε, πρέπει να τεθούν και είναι ε, αυτά τα ανοιχτή, ανοιχτοί λογαριασμοί. Η πρόεδρο, ναι, σα ευχαριστώ. 3 Μαΐου από τις 3 ε, έως 6.30 είναι η επόμενη συνεδρία τη Επιτροπής μας και συνεχίζεται και στις 4 ε, Μαΐου το πρωί, 9 με 12.30. Σας ευχαριστώ για την προσέλευση, ευχαριστούμε και τους διερμηνείς.